Good afternoon, my dear distinguished colleagues. Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, τον Επιτροπή κ. Φερχόικεν. Και το θέμα που έχουμε σήμερα στη διάταξη είναι η απόψε με τον κύριο Επίτροπο. Και θα ήθελα καταρχήν να του δώσω το λόγο να μας κάνει μια εισαγωγική παρουσίαση και μετά θα υπάρχουν κάποιες δυνατότητες αλληλής απόψεις. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω σήμερα πάλι μια δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων μαζί σας για διάφορα επίκαιρα θέματα και κάποια θέματα που προσβλέπουν ιδιαίτερα στο μέλλον. Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα έργο που πρέπει ακόμα να επιτελέσουμε από κοινού. Κατά τη γνώμη των γλυγορότερων δυνατών, δηλαδή το θέμα των φαρμακευτικών προϊόντων. που σας υπέβαλε η Κομισιόν τον Δεκέμβρη. Όλοι νομίζω εδώ στην αίθουσα γνωρίζουν ότι η φαρμακοβιομηχανία είναι από τους πιο δυναμικούς κλάδους ε, της Ευρώπης, ε, της ευρωπαϊκής οικονομίας και συμφωνούμε ότι πρόκειται για έναν ε, τομέα που θα αυξήσει ακόμα τη σημασία του και λόγω της δημοσιονομικής εξέλιξης αλλά και γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό θέμα για όλους. Ο, ξέρω ο καθένας όταν αρρώστησε πόσο σημαντική ήταν η υγεία του από εκεί και πέρα. Και στην Ευρώπη βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που όσο πάει και γυρνάει και γι' αυτό η υγεία θα είναι κοινωνικά ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ακόμη πιο σημαντικό στο μέλλον. Τα τελευταία χρόνια θετήσαμε μια σειρά σημαντικών νομοθετικών πράξεων που συμβάλλουν νομίζω σημαντικά στην βελτίωση της προστασίας της υγείας των πολιτών μας. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι νομίζω και το καταφέραμε να συνδέσουμε διάφορους στόχους και να τους συμβιβάσουμε μεταξύ τους. Και θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι <clears throat> όταν συζητάμε για διακανονισμού στον τομέα της ε, προστασίας της υγείας η υγεία και η ασφάλεια του ανθρώπου είναι το πρωτεύον θέμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία θέματα ανταγωνισμού, θέματα συμβατότητας με διεθνείς κανόνες, θέματα μείωση της γραφειοκρατίας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Αλλά όταν συζητάμε για θέματα υγείας, η ασφάλεια και η προστασία της υγείας είναι τα πρωτεύοντα θέματα, ο πρωτεύον στόχος. Έχουμε υιοθετήσει τέσσερις σημαντικές νομοθετικές πράξεις που νομίζω ότι πληρούν τους όρους αυτούς. Φαρμακευτικά διασκευάσματα για τα παιδιά, σύγχρονες θεραπείες, βελτιωμένες διατάξεις για την έγκριση ε, φαρμάκων και ε, κανόνες που αφορούν με τα κατάλοιπα φαρμακολογικά ενεργών ουσιών στην παραγωγή τροφίμων. Δεν αρκούμεθα σε αυτά όμως. Έχουμε μπροστά μας ακόμα τις προτάσεις που είπε η Κομισιόν το Δεκέμβριο. Πρόκειται για μια πρόταση που αποτελείται από τέσσερα τμήματα, μια πολιτική δήλωση, μετά νομοθετικές προτάσεις για την επιτήρηση των φαρμάκων, για τις ε, ε, και για την πλήρη ενημέρωση. Θα αναφερθώ στην παρατήρηση των προϊόντων αυτών. <clears throat> Για να είμαι ειλικρινής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν εκείνο που έγκαιρα επέστησε την προσοχή μου σε αυτό το θέμα, το τόσο σημαντικό. Συζητήσεις που είχαμε εδώ στο σώμα και που έπεσαν πολύ νωρί την προσοχή μου στο γεγονός ότι υπάρχει εδώ ένα σημαντικότατο πρόβλημα όχι για την Ευρώπη αλλά που μπορεί να καταστεί δραματικό και στην Ευρώπη εάν δεν δράσουμε. Και μου φάνηκε ότι ήταν καλύτερα να δράσουμε το γλυγορότερο δυνατόν και να μην περιμένουμε να έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δραματική κατάσταση και στη βιασύνη μας μετά ίσως να μην αντιδράσουμε σωστά. στην Ευρώπη δεν, θεωρούν πολύ ότι δεν υπάρχει ένα πρόβλημα με τα πλαστά αυτά φάρμακα. και ότι υπάρχουν μόνο στις πωλήσει μέσω διαδικτύου. Αυτό δεν είναι σωστό. Έχω να σας πω ότι το 2005 στα εξωτερικά μας σύνορα πράγμα που δεν είχε καμία σχέση με αγορές διαδικτύου και online κλπ. Από το 2005 έως το 2007 ή τα φάρμακα αυτά που μπορέσαμε να κατασχέσουμε στα σύνορα τετραπλασιάστηκαν σε όγκο. Σε πολλά τμήματα της ε, αλυσίδας εμπορίας βρέθηκαν αυτά τα φάρμακα. Και θέλω να σας πω ότι εάν κάπου σε ένα φαρμακείο βρούμε ένα πλαστό φάρμακο, αυτό σημαίνει ότι ανακαλούνται χιλιάδες συσκευασίε. Πράγμα που είναι πανάκριβο βέβαια. Κάθε μεμονωμένη λοιπόν ε, περίπτωση αφορά χιλιάδες συσκευασιών, άρα χιλιάδες ενδεχομένως ασθενών. Οι ασθενείς πρέπει να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στην ποιότητα των φαρμάκων που αγοράζουν νόμιμα. Και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε καθαρούς και σαφείς κανόνες για όλους σε όλα τα στάδια της εμπορίας και θα θέλουμε να είμαστε πιο αυστηροί στον έλεγχο των φαρμάκων, στην ε, εμπορία τράνζιτ και σε εξαγωγές και θα πρέπει επίσης να υπάρχουν ειδικά κα ε, στοιχεία ε, ασφαλείας στα φάρμακα τα οποία δίνονται μόνο με συνταγή παραδείγματος χάρη μία σφραγίδα φερρυπίν που αποδεικνύει στο καταναλωτή ότι αυτό η συσκευασία δεν έχει ανοιχτεί ακόμα. Και κάποιο χαρακτηριστικό δείγμα που να αποδεικνύει ότι αυτό που αναγράφεται στη συσκευασία είναι αυτό που είναι και μέσα στη συσκευασία και κάποια τεχνικά μέσα, κενό ή οτιδήποτε άλλο, βάσει του οποίου μπορεί κανένας να ε, παρακολουθήσει ακριβώς από πού ξεκίνησε η συσκευασία αυτή μέχρι να φτάσει στα χέρια του καταναλωτή. Και επίσης διάφορες διατάξεις για την επιτήρηση ασφάλειας των ε, ενεργών ουσιών. Θα ήθελα να σας πω κάτι για μια εκστρατεία περίεργη κάπως κατά τη διάρκεια των μελέτης ε, των διατάξεων αυτών, όπου το ότι υπάρχει η πρόθεση κάποια συγκεκριμένη δυνατότητα εμπορίας να απαγορευτεί, το λεγόμενο παράλληλο εμπόριο, αλλά αυτή δεν ήταν η πρόθεση, γιατί παράλληλο εμπόριο είναι κατά μιας απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μία οικονομική δραστηριότητα που επιτρέπεται ρητά στην εσωτερική αγορά. Δεν πρέπει να αλλάξουμε, αλλά από την άλλη μεριά είναι σαφές ότι για το παράλληλο εμπόριο όσον αφορά την ασφάλεια των ε, φαρμακευτικών πάντα θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες όπως και για τις άλλες οδούς εμπορίας. Όχι περισσότερο και όχι λιγότερο. Δεν προτιμάμε κανέναν, δεν επιβάλλουμε ιδιαίτερο βάρος σε κανέναν. Όσον αφορά τις ε, νομικές ε, διατάξεις για την επιτήρηση των φαρμάκων, πρόκειται για διατάξεις επιτήρησης των φαρμάκων που έχουν ήδη επιτραπεί να κυκλοφορούν. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο θέμα, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι για ε, φάρμακα που έχουν ήδη εγκριθεί, παρόλε σε ε, αυστηρές διατάξεις υπάρχουν πλαστά φάρμακα στην αγορά. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε μια μεθόδο σύμφωνα με την οποία γλίγορα και αποτελεσματικά να γίνεται γνωστό παντού και να μπορούν να υιοθετηθούν τα απαραίτητα μέτρα. Οι παραγωγοί δηλαδή, θα πρέπει να εισαγάγουν ένα αποτελεσματικό σύστημα επιτήρησης θα πρέπει να έχουν και ένα σύστημα για να ε, μπορούν να ενημερώσουν για άγνωστες μέχρι τούδε και αρνητικές ε, επιπτώσεις. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να μπορεί ο καταναλωτής όταν αισθάνεται κάποια παρενέργεια, έχει την εντύπωση ότι κάποιο φάρμακο δεν του κάνει καλό, να μπορεί να μην είναι ένας ε, απλώς παθητικός ασθενής αν θέλετε, αλλά ένας ασθενής που αντιδρά σε αυτό και που δηλώνει όπου πρέπει να δηλωθεί η παρενέργεια αυτή. Και θα φτάνουμε βέβαια στο θέμα της ε, βελτιωμένης ενημέρωσης του ασθενούς. Αυτό είναι δύσκολο θέμα το είχαμε συζητήσει ήδη αναλυτικά στην ακρόαση τέλη του 2004 με είχατε υποχρεώσει να υποβάλω μια σχετική πρόταση η οποία υπάρχει τώρα επιτάπητος. Και θα ήθελα να σας αναπτύξω για άλλη μια φορά το σημείο κίνησης της σκέψης μου. Ο στόχος είναι ο ασθενής και τα δικαιώματά του να τεθούν στο επίκεντρο των σκέψεών μας. Όλα όσα σχετίζονται με υγεία θα πρέπει να προσανατολίζονται στον ασθενή, στον άνθρωπο. Είπα ήδη ότι το... η υγεία είναι το ύψιστο αγαθό όλων μας. Και η ανάγκη να είμαστε πλήρως επνήμεροι για όλα που σχετίζονται με την υγεία μας αυξάνεται συνεχώς στην κοινωνία μας. Και η προσφορά πληροφοριών επίσης ευρύνεται. Αυτό είναι και επακόλουθο των ε, σύγχρονων μέσων πληροφορίας και ενημέρωσης. Όταν είναι κανένας online στο διαδίκτυο και ξέρει αγγλικά έχει ε, πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορίες χωρίς να ξέρει πάνωτε... ποια είναι η πηγή της πληροφορίας αυτής και πόσο σοβαρά πρέπει να πάρει υπόψη του τις πληροφορίες που διαβάζει. Ξέρω ότι η ενημέρωση των ασθενών είναι ένα φιλεγόμενο θέμα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω όμως μια βασική αρχή κάθε δημοκρατίας. Σε μια δημοκρατία δεν ε, χρειάζεται αιτιολόγηση για την ενημέρωση των πολιτών. Όχι. Στη δημοκρατία πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση εάν δεν υπάρχει ενημέρωση των πολιτών. Αυτό μου φαίνεται είναι πάρα πολύ κεντρικό θέμα. Και μέχρι στιγμής απορούσα πολλές φορές στην συζήτηση αυτή που μου ζητούσε να αιτιολογήσω γιατί θέλω να ενημερώσω τον ασθενή. Και λέω, και γιατί πρέπει να αφήσουμε τον ασθενή να μην ξέρει αυτά που θα μπορούσε να μάθει. Λοιπόν, οι ασθενείς χρειάζονται πληροφορίες. Κυρίες και κύριοι ε, βουλευτές, ο καθένας στην οικογένειά του, μεταξύ των φίλων, των συνεργατών, συναδέλφων ή και ο ίδιος, το έχει ζήσει αυτό πολύ σοβαρά. όποιος επλήγει, ο ίδιος ή κάποιος που γνωρίζει με μια βαριά ασθένεια, πραγματικά βαριά ασθένεια, και οι ελπίδες είναι μικρές. Οι θεραπείες που υπάρχουν να μπορούν να οδηγήσουν στην ίαση, μπορείτε να είστε σίγουρες. Ή ο άμεσα ενδιαφερόμενος ή το περιβάλλον όλοι αυτοί που τον αγαπούν, κάνουν τα πάντα για να δουν μήπως υπάρχει ίσως κάποια ευκαιρία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι. Και αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένω. Και αυτό που μας λένε και οι, οι γιατροί στην πράξη, ότι έρχονται κάποιοι και λένε «Ε, εδώ κάτι βρήκα, υπάρχει αυτό το φάρμακο, γιατί δεν μου το δεν μου δίνετε μια συνταγή γι' αυτό. Υπάρχει μια θεραπεία δεν μπορώ να την ακολουθήσω. Και δεν είναι πάντα πολύ εύκολο να εξηγήσει κανένα γιατί η θεραπεία αυτή έχει πάρα πολλέ παρενέργειε, δεν είναι ακόμα καλά ελεγμένη. Αλλά υπάρχει ανάγκη ενημέρωση. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το status quo που έχουμε σήμερα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών να έχουν υψηλής ποιότητα πληροφορίας. γιατί εκείνοι που είναι πιο μορφωμένοι ίσως και έχουν πρόσβαση έχουν οι περισσότερες πληροφορίες. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να δώσουμε τις πληροφορίες σε εκείνους που τις χρειάζονται άμεσα. Δηλαδή στους πιο ηλικιαμένους στην κοινωνία μας που έχουν τις περισσότερες ανάγκες ενημέρωσης για την υγεία τους. Πριν από μερικές μέρες διάβασα μια συνέντευξη τύπου ενός μέλους του σώματος στην οποία ανισχυρίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή θέλει να μην είναι πια τόσο αυστηρή, ε, αυστηρές οι διατάξεις ε, διαφήμισης φαρμάκων που δίνονται μόνο με συνταγές. Δεν συζητιέται το θέμα, σας το λέω ξεκάθαρα. Τα φάρμακα αυτά δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται. Απ' την άλλη μεριά δεν συμφωνώ με οποιονδήποτε λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση μεταξύ διαφήμισης και πληροφορίας. Φυσικά υπάρχει διαφορά. Κάθε δημοσιογράφος Βρυξέλλης εδώ το αποδεικνύει καθημερινά ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ πληροφορίας και διαφήμισης. Κάθε βουλευτής το αποδεικνύει αυτό. Και γι' αυτό, μετά από τις σκέψεις αυτές, η Κομισιόν έκανε τις αρχικές προτάσεις. Να είναι ελεύθερη η πληροφόρηση και η ενημέρωση. Πώς θα γίνει αυτό μόνο ορισμένες πληροφορίες επιτρέπεται να δοθούν ελεύθερα, δηλαδή εκείνες που έχουν ήδη εξεταστεί από τις αρχές και που αναφέρονται στα, στα χαρτάκια που συνοδεύουν τα φάρμακα. Υπάρχουν ναι, πολλές μελέτες που έγιναν στη Μεγάλη Βρετανία και που αξιολόγησε η ΕΜΕΑ, η υπηρεσία αυτή, η δική μας υπηρεσία που είναι στη Μεγάλη Βρετανία και βάσει αυτών των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης άλλαξε η ΕΜΕΑ την στάση της για την ενημέρωση των ασθενών. Οι μελέτες αυτές αποδεικνύουν ότι 5% όλων των ο, ο, όλης της ε, νοσήλευσης νοσοκομεία ασθενών οφείλεται στο γεγονός κακής χρήσης των φαρμάκων θα μπορούσαν να αποφευθούν το 5% αυτών των, ε, <clears throat> των περιπτώσεων εάν ήταν καλύτερα ενημερωμένοι οι ασθενείς. Πολλοί λένε βέβαια ότι θα πρέπει εδώ να είμαστε προσεκτικοί γιατί αν οι ασθενείς έχουν όλες αυτές τις πληροφορίες αυτό ίσως αυξήσει το κόστος στον ε, υγειονομικό τομέα γιατί θα ζητάνε κάποια ακριβά φάρμακα τα οποία δεν θέλουμε να τους δώσουμε. Αυτό το επιχείρημα δεν στέκεται. Γιατί ακριβώς αυτές οι μελέτες αποδεικνύουν ότι ο ενημερωμένος ασθενής δεν είναι πιο ακριβώς ασθενής όπως θεωρούν πολλοί, αλλά τον αντίον συμβάλλει στη μείωση του κόστους της ε, υγειονομικής περίθαλψης. Δεύτερον, οι πληροφορίες στις οποίες αναφέρομαι ε, επιτρέπεται να δίνονται στο διαδίκτυο μόνο ή σε γραπτές ερωτήσεις, σε, σε, σε γραπτές απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις ή σε κάποιες δημοσιεύσεις που σχετίζονται με θέματα της υγείας. Το ποιες είναι οι δημοσιεύσεις αυτές που ζητήσουν με θέματα της υγείας είναι θέμα που θα αφήσουμε ελεύθερα στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν. Θα μπορούν βέβαια να είναι κάποιες δημοσιεύσεις του κλάδου που αφορούν μόνο ε, ιατρικές δημοσιεύσεις αλλά θα μπορούσε και κάποια συγκεκριμένη εφημερίδα ή περιοδικό που έχει ένα τμήμα που αφορά θέματα υγείας θα πρέπει να είναι δυνατόν εκεί να δημοσιεύονται αυτές οι πληροφορίες. Και σας λέω, η, την ακριβή διάκριση ποιε είναι αυτές οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να γίνει από τα κράτη-μέλη. Οπωσδήποτε οι δημοσιεύσει αυτές θα πρέπει να τηρούν πολύ αυστηρά κριτήρια ποιότητας και επίσης τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν αποτελεσματικού μηχανισμούς ελέγχου. Ο όλοχο αυτός θα πρέπει να γίνεται καταρχήν πριν από τη δημοσίευση. Μέσα στα πλαίσια σχετικά αποτελεσματικών συστημάτων που υπάρχουν ήδη σε ορισμένα κράτη-μέλη. Δηλαδή έλεγχος ex μπορεί να επιτραπεί μόνο στην περίπτωση κατά οποία υπάρχει ήδη ένα σύστημα που προσφέρει αρκετέ αρκετές εγγύσεις για τους ελέγχους εξάντε. Αυτή είναι η πρόταση για το θέμα αυτό και θα ήθελα να πιστήσω και την προσοχή σας ότι στην ανακοίνωση της ε, Κομισιόν υπάρχουν και διάφορα άλλα θέματα πολύ μεγάλη σημασία. Παραδείγματος χάρη διεθνής συνεργασία μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για να εξασφαλιστεί η αναγνωστικότητα της φαρμακευτικής μας βιομηχανίας και να εγγυηθούμε την ασφάλεια των φαρμάκων στην ε, ευρωπαϊκή αγορά. Η ανακοίνωση αυτή αναφέρει ξεκάθαρα ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα που θα πρέπει να αναλυφθούν για να μπορέσουν να προωθηθούν τα αποτελέσματα του λεγόμενου φόρουμ φαρμάκων. Είμαι γνώμη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ γλίγορα όρισε τους συζητητές για τα μεμονωμένα τμήματα της δέσμης αυτής. Είχα ήδη την ευκαιρία να, να συζητήσω με τους περισσότερους, όπως πάντα η Κομισιόν προσφέρει την πλήρη υποστήριξή σας, υποστήριξή της συγγνώμη για την εργασία σας και ελπίζω ότι η δέσμη αυτή θα μπορέσει να προωθηθεί γλίγορα προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης. Έρχομαι στο δεύτερο θέμα, το οποίο σχετίζεται, είναι γειτονικό κατά κάποιο τρόπο, τα καλλιντικά. Στα πλαίσια της βελτίωσης και απλοποίησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας υποβάλλουμε πρόταση για τον τομέα των καλλιντικών, στην οποία πρώτα συγχωνεύονται 55 διαφορετικά νομοθετικά κείμενα μειώνοντας έτσι περίπου και κατά 50% το κόστος της σχετιζόμενης με τα κείμενα αυτά γραφειοκρατίας. Έχουμε προχωρήσει στο μεταξύ με το θέμα αυτό στην διαβούλευση και είμαι ικανοποιημένο διότι Συμβούλιο και Κοινοβούλιο προσεγγίζουν άλληλα. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο όπως είπα για το γεγονός αυτό και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε πρώτη ανάγνωση πριν λήξει η θητεία του παρόντος Κοινοβουλίου. Εάν τα βλέπω καλά τα πράγματα φαίνεται να μένει ένα δυσχερές θέμα πώς δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε, πώς θα χειριστούμε ορισμένα υλικά συστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή καλλιντικών προβλέπεται ε, ανακοίνωση για ορισμένα κοινοποίηση μάλλον για ορισμένα από τα συστατικά αυτά. Προτιμώ να μην δεσμευτώ σήμερα εν ώψη και του τριμερούς διαλόγου. Ε, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα όπως είπα να προωθηθεί μια λύση. Η Επιτροπή θα κάνει τη δική της προσπάθεια να συμβάλλει στην επίτευξη λύσης. Εγώ ήδη έχω προτείνει να συζητήσω με τους εισηγητές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως θα πράξει πάντο δυνατόν για να συμβάλλει στην επίλυση του εναπομένοντος θέματος. Σε ό,τι αφορά τώρα τα νάνο υλικά αυτά, περί των οποίων στην ουσία πρόκειται, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και σε άλλους τομείς. προσπαθούμε να θεμελιώσουμε τις ρυθμίσεις μας σε αυστηρά επιστημονική βάση. Science-based regulation. Αυτό απαιτεί και η διεθνής πρακτική. Δεν είναι όμως και πάντοτε τα συμπεράσματα της επιστήμης απόλυτα σαφή και μονοσήμαντα. Καμιά φορά μάλιστα εμφανίζονται και αντιφατικά. Πρόσφατα μάλιστα συνέβη αυτό δύο φορές σε ένα δύσκολο και σημαντικό θέμα των χημικών ουσιών σε παιχνίδια για παιδιά και επίσης στο θέμα της αντιμετώπισης του εισαγόμενου κρέας πουλερικών το οποίο ε, είχε γίνει αντικείμενο Επεξεργασία με ορισμένα αντιβακτηριδιακά προϊόντα, χλώριο στην ουσία. Ε, εδώ η επιστήμη μας έδωσε αντιφατικά συμπεράσματα. Για τα νάνο ε, προϊόντα αυτά, για τα νάνο υλικά, συμβαίνει ορισμένε φορέ το ίδιο. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να εντείνουμε τι προσπάθειέ μα ώστε να εμβαθύνουμε τη γνώση μα για τι συνέπειε αυτών των υλικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το πράξει αυτό θα ενισχύσουμε λοιπόν, θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να έχουμε μια στέρεα επιστημονική βάση για την χρήση αυτών των νάνο υλικών και βεβαίως θα ενημερώνουμε τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις προόδους ώστε να μπορούν να συνάγονται και τα απαραίτητα συμπεράσματα. Συμφωνώ απολύτως. Εάν αποδειχθεί από την εργασία αυτή ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι τους οποίους δεν προβλέψαμε θα πρέπει τότε να προβούμε σε κάποιες δράσεις με μεγάλη ταχύτητα. Μπορεί να ε, αποδειχθεί και το αντίθετο, ότι αναμένουμε κινδύνους εκεί όπου δεν υπάρχουν. Και πάλι θα πρέπει να αλλάξουμε τη στάση μας. Όμως, το θέμα αυτό ότι θα κάνουμε ακριβώς με τα ανανοηλικά σε αυτήν την προκείμενη πρόταση οδηγίας, θα το συζητήσω με τους εισηγητές, με λεπτομέρεια και γνωρίζοντας ποια είναι η πρόοδος των διαβουλεύσεων με το Συμβούλιο, Κοινοβουλίο Συμβουλίου. Το ίδιο και για, την, ε, για τα πλαστά ε, καλλιντικά. Καλλιντικά τα οποία μετά ε, βάζουν οι άνθρωποι πάνω στην επιδερμίδα τους. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε την προστασία των καταναλωτριών και καταναλωτών απέναντι σε τέτοια πλαστά ε, καλλιντικά. Θα είναι σωστό να περιληφθεί και μια αιτηλογική σκέψη σχετικά με την οριζόντια νομοθεσία και ε, ρύθμιση για όλους τους παράγοντες μέσα στην αλυσίδα παραγωγής και προμήθειας και βεβαίως εποπτεία της αγοράς η οποία να διασφαλίζει ότι θα μπορούν να εντοπίζονται τα πλαστά υλικά και να παρακολουθούνται. Τελειώνοντας, επιθυμώ να θίξω ένα θέμα το οποίο υπερβαίνει και τα όρια της παρούσας ή επικείμενης νομοθεσίας και έχει κατά κάποιο τρόπο προγραμματικό χαρακτήρα για το επόμενο χρονικό διάστημα. Εν δηλαδή της οικονομικής κρίσης που μαστίζει όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να ε, ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο μαθαίνουμε όλοι ότι αυτή η άγωνη αντιπαράθεση μεταξύ οικονομίας και οικολογίας πρέπει να πάψει. Και ιδίως σε ό,τι αφορά την γνώση που αποκτούμε σιγά σιγά σχετικά <clears throat> με τις αλλαγές του κλίματος και τη δυνατότητα της Ευρώπης να αποτελέσει υπόδειγμα για τον αγώνα για την αντιμετώπιση των αλλαγών του κλίματος. Ο προβληματισμός αυτός είναι σαφές ότι υπερβαίνει τη, την προσπάθεια μείωσης μοναχά των ε, καυσαερίων, των αερίων του θερμοκηπίου. Να κάνουμε δηλαδή και ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας βιομηχανικής παραγωγής που να έχει χαρακτήρα αηφορίας. Στα αγγλικά θα το έλεγα και χωρίς καμία σύστολη, θα μιλούσα δηλαδή για μια πράσινη βιομηχανική επανάσταση. Επειδή όμως ε, μιλώ γερμανικά, ε, δεν τολμώ να χρησιμοποιήσω το επίθετο πράσινο, γιατί πράσινος στα γερμανικά έχει έντονα κομματικό χαρακτήρα. Πάντως ολόκληρη η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να ρίξει το βάρος της σε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί ενεργειακά αποδοτικά με κατά το δυνατόν περιορισμένη χρήση των φυσικών πόρων και φυσικά σε μια προσπάθεια να αναπτύξει διαδικασίες βιομηχανικής παραγωγής που να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον. Αυτά δεν χρειάζεται να τα θεμελιώσω οικολογικά, αυτό είναι αυτονόητο. Υπάρχει και οικονομική θεμελίωση. Για ποιο λόγο είναι σωστό να γίνει αυτή η προσπάθεια. μελλοντικές προοπτικές της ε, ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις παγκόσμιες αγορές θα βελτιωθούν εάν είμαστε σε θέση όχι μόνο να προσφέρουμε τεχνολογίες του περιβάλλοντος μόνο, γιατί ήδη είμαστε οι καλύτεροι σε αυτά, είναι δηλαδή κάποιοι τομείς της βιομηχανικής παραγωγής όπου δεν σημειώνεται κρίση η παραγωγή των τεχνολογιών ε, που είναι φιλικές με το περιβάλλον, αλλά και να προσφέρουμε και προϊόντα και τεχνολογίες που να επιτρέψουν και στους άλλους να βελτιώσουν την ε, προστασία του περιβάλλοντος από πλευράς τους. Για παράδειγμα, τα δομικά υλικά. Ούτε ιδέα έχουμε τι τρομερή βελτίωση μπορούμε να επιτύχουμε με τη χρήση δομικών υλικών που να έχουν οικολογικό χαρακτήρα. Ήδη στην Ευρωπαϊκή Αγορά προσφέρονται δομικά υλικά τα οποία επιτρέπουν την μείωση, τη δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση ενός κτίριου. Μπορούμε να φτιάξουμε ήδη σήμερα σπίτια και κτίρια, τα οποία όχι μόνο δεν απαιτούν ενέργεια για την θέρμανση ή την ψήξη τους, αλλά μάλιστα μπορούν και να παραγάγουν ενέργεια. Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για την Κίνα, για παράδειγμα αν με τον τρόπο αυτό ε, την βοηθήσουμε να λύσει το πρόβλημα της τεράστιας σπατάλης ενέργειας που προκαλείται από την χρήση εκεί δομικών υλικών τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη καθόλου τις ανάγκες του περιβάλλοντος. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο νομίζω είναι πιστικό. Τα αυτοκίνητα είναι άλλο παράδειγμα. Και ανεξαρτήτως της κρίσης που αντιμετωπίζουμε τώρα στην ευρωπαϊκή αυτοκίνητο βιομηχανία, γιατί βέβαια δεν είναι μόνο στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, σε όλη την αυτοκινητοβιομηχανία, παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, εμφανίζεται πλέον καθαρά ότι το αυτοκίνητο του μέλλοντος θα πρέπει να είναι ενεργειακά αποδοτικό. Και εφόσον η ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται τώρα σε μια φάση που κάπως δυσκολεύει η οικονομική κρίση, παρόλα αυτά, ε, όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η φάση αναπροσαρμογής, θα κρατήσει ακόμα μερικά χρόνια, τότε οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές θα έχουν πραγματικά πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας στην παγκόσμια αγορά να μπορούν να προσφέρουν δηλαδή το αυτοκίνητο του μέλλοντος. Και θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα πολλά παραδείγματα. Πέρσι σας είχα υποβάλει πρόταση ενός σχεδίου δράσεως για μια αηφόρο βιομηχανική πολιτική που ε, θα ήταν ε, μια δέσμη μέτρων που ε, συμπληρώνει την πολιτική του περιβάλλοντος που έχει ήδη εγκρίνει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με την ανάπτυξη νέων συνθήκων πλαισίων για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και για την βελτίωση των προϊόντων της. Εκτός αυτού έχουμε σκοπό να εκμεταλλευτούμε και τις δυνάμεις της αγοράς. Δηλαδή να τονώσουμε την πλευρά της ζήτησης, να αναπτυχθεί μια ζήτηση για περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι ενήμερος ο καταναλωτής, διότι μόνο ο ενημερωμένος καταναλωτής θα ενδιαφερθεί για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα για αποδοτικότητα του προϊόντος. Και είμαι βέβαιος ότι εάν τα καταφέρουμε σωστά, οι καταναλωτές θα είναι και οι καλύτεροι μας σύμμαχοι για να επιτύχουμε αυτή την, αυτόν τον αναπροσανατολισμό που απαιτείται. Η Επιτροπή σας έχει παίξει σημαντικό ρόλο ήδη τον Απρίλιο του 2005 με την ε, οδηγία Eco Design που ήταν ένα παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης ενοποιημένης πολιτικής στην Ευρώπη γιατί καλύπτει το προϊόν σε ολόκληρο τον κύκλο της ύπαρξής του για όλα τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και είναι έτσι και σημαντική συμβολή της στην προσπάθεια μείωσης του διοξιδιού του άνθρακος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τώρα να επεκταθεί αυτή η οδηγία και να περιληφθούν όλα τα προϊόντα τα οποία έχουν κάποια σχέση με την ενέργεια. Όχι μόνο δηλαδή εκείνα τα οποία καταναλώνουν άμεσα ενέργεια, αλλά οποίον και των οποίων η χρήση έχει κάποια συνέπεια στην ενέργεια. Φαίνω παράδειγμα, δομικά υλικά, παράθυρα, ε, αυτά τα τηλέφωνα του ντους. Υπάρχουν ατελείωτα παραδείγματα που μπορεί κανείς να αναφέρει εν προκειμένου που έχουν δηλαδή κάποια αποτελέσματα στην κατανάλωση ενέργειας. Επί του παρόντος μου φαίνεται σημαντικό να ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος στα προϊόντα εκείνα όπου μπορούμε γρήγορα να επιτύχουμε κάποια αποτελέσματα στην ε, κατανάλωση ενέργειας και επομένως στο περιβάλλον. Είμαι όμως βέβαιος ότι μέσω και μακροπρόθεσμα θα πρέπει να βελτιωθεί η ε, ενεργειακή αποδοτικότητα και η φιλικότητα προς το περιβάλλον, η οικολογικότητα δηλαδή όλων των ευρωπαϊκών προϊόντων και είμαι πεπισμένος ότι και αυτή εδώ η οδηγία θα μπορέσει να τεθεί σύντομα σε ισχύ και είμαι βέβαιος ότι τα σχετικά βήματα για μια, μια πιο αποδοτική σε χρήση ενέργειας παραγωγή θα μπορέσει και αυτή και να καταστεί δυνατή. Και αυτά που σας είπα τώρα μόλις αποτελούν στην ουσία ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο βέβαια δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί ούτε πλέον στη διάρκεια της θητείας της παρούσας επιτροπής ούτε και του παρόντος κοινοβουλίου. Δίνει ωστόσο μια κατεύθυνση, ένα προσανατολισμό για τις ενέργειες που θα πρέπει να αναλάβει το Κοινοβούλιο στην επόμενη θητεία του, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δική της επόμενη θητεία. Εν τω μεταξύ, στα τελευταία χρόνια, με ορισμένες πραγματικά μοναδικές παγκόσμια προτάσεις έχουμε καταφέρει να βάλουμε κάποιες κατευθύνσεις αλλά και να συλλέξουμε κάποιες εμπειρίες και παρακαλώ μην ακούτε εκείνους που λένε ότι τώρα βρισκόμαστε πια αποτελματωμένοι μέσα στην κρίση, ας τα ξεχάσουμε όλα αυτά τα ευγενή περί περιβάλλοντος και ε, τα σχετικά και ας φροντίσουμε να ξυπνήσει και πάλι η κατανάλωση των νοικοκυριών. Βεβαίω και εγώ θέλω να τονωθεί και πάλι η ζήτηση. Δεν υπάρχει όμως κανένας λόγος να πούμε ότι δεν χρειάζεται ταυτόχρονα να τονώσουμε την ζήτηση υπέρ οικολογικών και ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. Θεωρώ μάλιστα σωστό μέσα στην κρίση να φροντίσουμε ώστε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που πρέπει να λάβουμε για την αντιμετώπιση της κρίσης να μην θέσουν σε κίνδυνο τους μακροπρόθεσμους ή και μεσοπρόθεσμους στόχους μας. Θεωρώ λοιπόν ότι μια αηφόρος βιομηχανική πολιτική αποτελεί και το σωστό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much indeed. Uh, Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Επιτροπέ. 40 λεπτά προβλέπονται για την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο. Έχω ήδη σημειώσει 10 ομιλητές. Θα σας διαβάσω τον κατάλογο για να τον ολοκληρώσουμε. Bois, Dagmar Parent, Mr. Adamo, Christina Klaas, Peter Lise, Gutierrez Cortines, Mr. Kramer, McEwan, Thomas Sulmer, Harold Doyle. Is it all? Anders Wickman will be added to the list. Kathy Sinot will be added to the list. Προσθέτουμε και την Kathy Sinot. Άλλος κανείς? Όχι, οπότε ολοκληρώνεται ο κατάλογος με τους αγορητές. Ο συνήθως θα δώσω πρώτα το λόγο σε τέσσερα μέλη. Για τον πρώτο γύρο ερωτήσεων θα δώσω τον λόγο στον Επίτροπο να απαντήσει και ούτω καθεξής. Ο Τζον Μπάουις έχει το λόγο πρώτα. Ευχαριστώ τον κύριο Βερχόγγεν για την ευρία αυτή επισκόπηση που μας έκανε και μάλιστα επεκτάθηκε σε πιο απότερο χρονικό ορίζοντα μετά τις εκλογές και μετά το πέρας της θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο θέματα. Το ένα αφορά τη μνήα σε κτίρια αποδοτικά από άποψη ενέργειας, αλλά και σε ενεργειακά αποδοτικά αγαθά και υπηρεσίες. Συμφωνώ μαζί σας ότι αυτή θα πρέπει να είναι η βασική μας κατεύθυνση. Ερωτώ όμως, τι κάνουμε για να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο, όχι μόνο νομοθετικά, αλλά και με την πολιτική μας για τις, κρατικές προ... για τις προμήθειες γενικώ. <clears throat> το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχουν μεγάλη ισχύ στις προμήθειες. Αν το χρησιμοποιήσουν αυτό το δικαίωμα που έχουν, στα κτίρια που αγοράζουν, στις υπηρεσίες, ε, αλλά και άλλοι οργανισμοί όπως η ΕΤΕ, η ΕΚΟ κτλ. Αν χρησιμοποιήσουν αυτή την εξουσία που έχουμε σε θέματα προμηθειών, προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι μπορούμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο. Επανέρχομαι τώρα στη δέσμη των φαρμακευτικών προϊόντων. Συμφωνώ σε γενικέ γραμμέ με τον Επίτροπο. Θα ήθελα πάντω να υπάρξει ένα σωστό συντονισμό μεταξύ των γενικών διευθύνσεων για τα θέματα αυτά. Γιατί το θέμα τη ασφάλεια των ασθενών, που είναι συναφές με την διασυνοριακή υγεία. Έχουμε το θέμα της εποπτείας για τα φάρμακα, που επίσης έχει μια πτυχή ε, προστασία των ασθενών. Έχουμε ε, τα τραυματισμούς από σύριγγες, ε, θέμα του σπίτλ. Έχουμε τα νοθευμένα φάρμακα, τα πλαστά φάρμακα αναφέρθηκε, που εμπίπτει σε άλλη γενική διεύθυνση, το χαρτοφυλάκιο της κυρίας Βασιλείου για ανθιγυνά επαγγέλματα. Πώς μπορούμε λοιπόν να συντονίσουμε τις διάφορες διευθύνσεις της Επιτροπής ώστε να υπάρχει μια οριζόντια πτυχή, για παράδειγμα, της ασφάλειας των ασθενών σε όλες τις πολιτικές. Η ενημέρωση επίσης των ασθενών είναι κάτι που επιθυμούν διακαώσει οι ομάδες των ασθενών. Αλλά ε, θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης, γιατί δεν θέλουν διαφήμιση, θέλουν ενημέρωση. Υπάρχει όμως μια φαιά ζώνη μεταξύ των δύο. Αυτό το, της έμεσης διαφήμισης, της διαφήμιση, διαφήμισης, της προβολής προϊόντων με έμεσο τρόπο. Εκεί μήπως δημιουργηθεί ένα παραθυράκι, για παράδειγμα, μήπως θα μπορούν κάποιες τηλεσυρές ή ε, ραδιοφωνικές σειρές να έχουν μέσα στο κείμενο της τηλεοπτικής σειράς τη μία ενός προϊόντος, το, το σήμα ενός προϊόντος στη μάρκα, οπότε έμεσα προβάλλεται αυτό προς τον ακροατή ή θεατή. Είναι ένα είδος διαφήμιση. Έμεση μεν, διαφήμιση δε. Αυτό θα πρέπει να αποσαφινιστεί κατά τη γνώμη μου. Σας ευχαριστώ. Η Ντάγμα Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ωραίο ότι βρισκόστε έτσι σε φόρμα και έχω κάποιες παρατηρήσεις για τη δέσμη για τα φαρμακευτικά προϊόντα αλλά και για τα καλλινικά. Συμφωνώ τα μαζί σας ότι οι γραμμές συζήτησης είναι πληκτικές για ορισμένες προτάσεις. Δεν καταλαβαίνω ότι όσον αφορά τα πλαστά ε, φαρμακά, ένα πραγματικά κίνδυνο ε, προϊόν, συζητιέται καταρχήν κατά πόσο επιτρέπεται ή όχι το παράλληλο εμπόριο. Ούτε καταλαβαίνω γιατί η δεύτερη σκέψη ορισμένα κράτη-μέλη είναι ότι ίσως αυτό ε, οδηγεί σε αύξηση του κόστους ε, της δημόσιας υγείας. Όταν μιλάμε για ε, κάποια φάρμακα που μπορούν να αποφύγουν μια θρόμβωση παραδείγματος χάνει και το, παίρνει ο ασθενής ένα φλαστό φάρμακο που οδηγεί ή που επιτρέπει τη θρόμβωση και πεθαίνει. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, που πρέπει να πάρουμε μέτρα τα οποία πραγματικά αποκλείουν κάτω το δυνατόν την, ε, ε, τα πλαστά αυτά φάρμακα. Εγώ ως πολιτική, ε, ως πολιτικός μου ζητούνται να έχω ε, ευφυείς λύσεις για διάφορα πράγματα. Εγώ το ίδιο περιμένω και από εκείνους που δρούν στον επαγγελματικό κόσμο που θα πρέπει να ορίσουν το πλαίσιο για να είναι κατά δυνατόν αδύνατες ή η αδύνατη πλαστοποίηση των ε, φαρμάκων αυτών. Κάτι που με ενοχλεί σχεδόν ακόμα περισσότερο όσον αφορά τα πλαστά ε, φάρμακα όσο η περί της σχεδόν συζήτηση για, την, ε, το παράλληλο εμπόριο είναι τα πλαστά, οι πλαστές ενεργές ουσίες. Γιατί αυτό παράγεται συνήθως σε κάποια γκαράζ, ας πούμε, σε κάποια μικροεργαστήρια, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδηγούν σε πάρα πολύ αποδοτικό εμπόριο. Και εκεί να σταματήσουμε, εκεί να ε, διακόψουν να κατανοήσουμε έγκαιρο ότι γίνεται αυτή η παροχή πλαστών ενεργών ουσιών. Δεν βρήκα καμία απάντηση κύριε Επίτροπε που να με ικανοποιεί εμένα, ούτε άκουσα καμία απάντηση από οποιοδήποτε άλλο. Ίσως έχετε κάποιες καλές ιδέες εσείς. Ενημέρωση των ασθενών τώρα. Ένα θέμα που με έχει απασχολήσει και πρωτού έρθω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, ε, ε, ένας τρόπος προστασίας αυτών των πολύ ασθενών μελών της κοινωνίας μας. Πολλά κάναμε, πολλά θετικά κάναμε, αλλά η ενημέρωση των ασθενών, η ενημέρωσή τους δηλαδή όσον αφορά τη θεραπεία μιας ασθένειας, είναι κάτι που θα πρέπει επίσης να πραγματοποιείται. Και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ξεκάθαρα ότι αυτή η πληροφορία δεν είναι μόνο πληροφορία για κάποιο φάρμακο και για άλλα πράγματα. Δηλαδή, εάν κάποιος έχει μια πολύ βαριά ασθένεια και πρέπει να παίρνει φάρμακα με παρενέργειες, πρέπει να ξέρει ποιες είναι οι δυνατότητες να αλαφρύνουν οι παρενέργειες αυτές. Ποιε είναι οι δυνατότητε για να αποφευθούν κάποιε ψυχολογικέ παρενέργειε, παραδείγματο χάρη. Και δεν θέλω κανένα να τον υποχρεώσω να πάει να δει μία ιστοσελίδα αμερικανική. Ξέρω τι σημαίνει να έχει κανένας ενημέρωση για μια δύσκολη ασθένεια. Εγώ θεωρώ ότι είμαι και εφής και σε θέση να χειριστώ το διαδίκτυο. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν εύκολο ούτε και για μένα να έχω τις πληροφορίες αυτές. Όποιος μπορεί δηλαδή να απλουστεύσει Ε, τα πράγματα και να λέει ότι αυτό είναι μονάχα μια εύκολη λύση για τους παραγωγούς, δεν έχει καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Στα λίγα λεπτά που μου αποβαίνουν κύριε Επίτροπε θέλω να αναφερθώ στα καλλιντικά. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την συνεργασία με τις υπηρεσίες γενικής σας διεύθυνσης που με σαφήνεια ε, πρόθεσαν αυτά που και εμείς όλοι τα θεωρούμε σημαντικά και είμαι ευγνώμων που για την νανοτεχνολογία μπορούμε τώρα να δούμε ποια είναι τα προβλήματα. Ελπίζω να τα κατάλαβα. Δεν θέλω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεωρηθεί ότι είναι εχθρικό προς τεχνολογία ή προς την πρόοδο. Και είμαι σίγουρη ότι οι γνώσεις μας για πολλές τεχνολογίες και για την τανακτορολογία πρέπει να αυξηθούν. Αλλά όταν συζητάμε κάτι που δεν το γνωρίζουμε πολύ καλά, όταν αναφερόμαστε σε ε, μικροσωματίδια ε, που τα φέρουμε στην επιδερμίνα και παιδιών ακόμα, θα πρέπει να εφαρμόσουν την αρχή της πρόληψης. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ότι για μας αυτή η αρχή της πρόληψης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αγαθό. Και γι' αυτό είμαι επιπισμένη ότι από κοινού και όσον αφορά την κοινοποίηση για τις τεχνολογίες αυτές και όσον αφορά την αδειοδότηση θα μπορέσουμε να βρούμε μια καλή λύση. Σήμερα το απόγευμα, όπως είπατε, είχαμε έναν ε, τριμερή διάλογο. Δεν συμφωνούμε σε όλα τα σημεία. Όλοι μαζί, ούτε η Κομισιόν με το Κοινοβούλιο, νομίζω θα μπορέσουμε να βρούμε έναν καλό συμβιβασμό. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed, uh, Mr. Σας ευχαριστούμε. Κύριος Αδάμου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τον ε, Επίτροπο Βερχόγγεν που ήρθε. Είμαι ο ε, για τα πλαστά φάρμακα, γι' αυτό και θα αναφερθώ κυρίως σε αυτό το θέμα. Το θέμα ε, των πλαστών φαρμάκων αφορά 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό, αυτός είναι ο τζίρος της βιομηχανίας πλαστών φαρμάκων. Η προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σωστή. Υπάρχουν όμω κάποιε αδυναμίε και λάθη που προσπαθώ να διορθώσω με τροπολογίε δικέ μου και των ε, συναδέλφων. Τι, ποια είναι καταρχήν αυτά τα πλαστά φάρμακα. Γιατί η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν περιλαμβάνει ορισμό των φαρμάκων προκειμένου να μην περιορίσει το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Εγώ το αντίθετο πιστεύω, ότι ένα ορισμό των φαρμάκων αυτών θα μα επιτρέψει να αναλάβουμε πιο έντονη δράση κατά των εγκληματιών. Γιατί η η μαφία των φαρμάκων είναι πραγματικά εγκληματική ενέργεια και θα πρέπει να ενισχύσουμε την διεθνή συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει να ξέρουμε τι ζητούμε, θα πρέπει να ξέρουμε το στοιχειώδες, τον ορισμό, τι, τι σημαίνει πλαστό φάρμακο. Και έχουμε και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας με ειδική ομάδα εργασίας για τα πλαστά φάρμακα. Εκεί, από εκεί θα μπορούσαμε να δανειστούμε έναν ορισμό που θα είναι διεθνώς αποδεκτός. Έρχομαι τώρα στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Όταν λέμε φαρμακευτικό προϊόν, τι εννοούμε. Ε, αναφέρεται η δραστική φαρμακευτική ουσία και το τελικό προϊόν. Βέβαια, ε, ο ε, ασθενής δεν καταναλώνει μόνο τη δραστική ουσία, αλλά και το περιτύλιγμα. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν επέκταση του πεδίου εφαρμογή τη οδηγία ώστε να καλυφθούν και φάρμακα που δίνονται χωρί συνταγή. Γιατί Ορισμένα φάρμακα υπόκειται στην υποχρέωση χορήγηση συνταγή σε ορισμένε χώρε, αλλά σε άλλε όχι. Οπότε για να είμαστε συνεπεί θα πρέπει να καλύψουμε όλα τα φάρμακα και αυτά που δεν συνταγογραφούνται. Τώρα έχουμε και το δούριο ύπο της, των πλαστών φαρμάκων. οι πωλήσει μέσω Ιντερνετ είναι ο η μεγαλύτερη πηγή ε, κέρδους για τους πολυδές πλαστών προϊόντων και όμως εκπίπτουν τις πρότασεις σε τέτοιου είδους ενέργειες. Θα πρέπει να περιλάβουμε και το ίντερνετ ε, σε αυτές τις ρυθμίσεις. Γιατί ένα μεγάλο τμήμα του λιανεμπορίου περνάει από εκεί. Σε ό,τι αφορά τις, ε, τις ετικέτες ή το, το σφράγισμα των φαρμάκων. Δεν υπάρχει πρόταση όμως για την εναρμόνιση της ασφάλειας στο μέλλον. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε την, τα πλαστά φάρμακα ε, συγκροτημένα και συνεπώς με ενίσχυση της συνεργασίας προκειμένου να εξαρθρώσουμε τα εγκληματικά κυκλώματα που δεν γνωρίζουν σύνορα. Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι διεθνείς προδιαγραφές μεταποίησης. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε ένα πιο αυστηρό σύστημα. Συμφωνώ με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα πρέπει όλοι να υπομισθούν με τις ευθύνες, οι φαρμακοβιομηχανοί, οι παρασκευαστές, οι χονδρέμποροι, όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας. Πάντως το κλειδί της επιτυχίας μας εδώ είναι η ευιστοποίηση, η συνειδητοποίηση του πολίτη. Γιατί όλο το έργο μας εδώ γίνεται πρώτα απ' όλα για τον καταναλωτή και τον ασθενή. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη δύο στοιχεία. Την ασφάλεια των ασθενών, να εξασφαλίσουμε να μην μετακυλίεται το κόστος στους καταναλωτές. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Σας ευχαριστώ. Και ο τέταρτος ε, ομιλητής, τέταρτη ομιλήτρια του πρώτου γύρου είναι η Κρίστα Κλάς. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Μία παρατήρηση όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα. Πληροφόρηση και διαφήμιση. Το, δεν είναι καθαρά οριοθυμένα αυτά. Υπάρχουν αυτές, ε, αυτά τα δικά περιοδικά περιοδικά που είπα είναι ειδικά για τα φάρμακα. Υπάρχουν ειδικά περιοδικά στα φαρμακεία στην Γερμανία παραδείγματος και ειδικά περιοδικά για τους γιατρούς. Καμιά φορά όμως εκεί λέγεται, γίνεται κάτι που είναι σαν διαφήμιση αλλά που είναι υποτίθεται για την ενημέρωση των γιατρών. Είναι δύσκολο να υιοθετήσουμε. Ε, εγώ ζήτησα το λόγο όταν αναφερθήκατε στην οδηγία για το eco-design και όποτε θέλει αυτό να διευρυνθεί σε άπειρα προϊόντα. Άπειρο με τρομάζει κύριε Επίτροπε. Γιατί είχαμε συζητήσει ότι δεν θέλουμε να βιαστούμε να υιοθετήσουμε κάτι τέτοιο και να δώσουμε επιταγή ελαφκό στην Εκτελεστική Επιτροπή δεν θέλω να ακολουθήσουμε την άκουσα αυτή. Θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι απαιτήσει για κάθε προϊόν. Υποθέτω ότι η αξιολόγηση κάθε προϊόντος θα είναι διαφορετική. Και θα πρέπει να ορίσουμε τι απαιτήσει αυτέ, τι ανάγκε αυτέ και γι' αυτό δεν θα πρέπει νομίζω πολύ ε, γλίγορα να προχωρήσουμε σε απειρά προϊόντα. Και θέλω να επιστήσω την προσοχή σας ότι και εμείς ως Κοινοβούλιο θέλουμε να μπορούμε να έχουμε λέγει και στα επιμέρους προϊόντα. Και θα πρέπει να το έχετε υπόψη σας αυτό όταν συζητάτε και το θέμα της αποτελεσματικότητας, γιατί θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ε, λήξης γιατί θέλουμε να αποσύρουμε τα φάρμακα αυτά <clears throat> από την αγορά, αλλά τα προϊόντα αυτά έχουν μία αξία ακόμα και δεν παραχθούν εκ νέου. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό να είναι παράγοντα που έχουμε υπόψη. Μας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, το λόγο έχει ο Επίτροπος. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Μπόις, σας παραπέμπω στην ανακοίνωση της Επιτροπής που συντάχθηκε ε, υπό, του, υπό την αιγίδα του Τσάρλι Μακρύβη για τις δημόσιες προμήθειες και που αναφέρει τα μέτρα που λαμβάνονται ε, στα πλαίσια της πολιτικής μας αυτής και μάλιστα ένας ολόκληρος αριθμός ε, ρυθμίσεων σχετικά με την προσπάθεια βελτιστοποίησης των δημοσίων προμηθειών ώστε να προτιμώνται οικολογικά εντό εισαγωγικών προϊόντα. Και ασχολούμεθα επί του παρόντος με ένα τέτοιο θέμα, ε, ιδιαίτερα επίκαιρο, ίσως ε, θα διαβάσατε ότι μας ανησυχεί ιδιαίτερα ο τομέας παραγωγής ε, οχημάτων που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίε κοινή ωφέλεια. Η παραγωγή ε, κανονικά μηνιαίως 40.000 40 τέτοιων οχημάτων. Τον Δεκέμβρη οι κατασκευαστές των οχημάτων αυτών έλαβαν 600 νέες παραγγελίες. Έχει καταρρεύσει πραγματικά η παραγωγή αυτή, έχει συμπαρασύρει και πολλές ε, θέσεις απασχόλησης. Μία δυνατότητα επανατόνωσης των, παραγωγή ε, της ε, παραγωγής αυτής θα ήταν οι χώρες μέλη να ζητήσουν από τις υπηρεσίες τους να προβούν σε αγορές οχημάτων χαμηλής κατανάλωσης και οικολογικού χαρακτήρα, εν πάση περιπτώσει, για παράδειγμα για τι δημόσιε μεταφορές. Όσον αφορά την ε, συνεκτικότητα της πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας απαντώ ότι το σύστημα του συλλογικού χαρακτήρα των αποφάσεων και της, της οργάνωσης δηλαδή της Κομισιόν σε βάση συλλογική, ακριβώς εκεί ε, σας αντιλέγει. Δηλαδή οι συνάδελφοι που έχουν καταρχήν την ευθύνη για ε, την υγεία έχουν συμμετάσχει σε όλες αυτές τις, απόψεις, τις αποφάσεις. Εάν τώρα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει την πρόθεση να αλλάξει την κατανομή των χαρτοφυλακίων εντός της Κομισιόν, αυτό δεν το γνωρίζω, ούτε άλλωστε μου αρμόζει να εκφραστώ επ' αυτού. Οι δικές μου εμπειρίες, όντας πλέον για 10 χρόνια επίτροπος, είναι ότι το σύστημα που έχουμε εξασφαλίζει επαρκώς την λήψη υπόψη όλων των πτυχών ε, κατά την εκπόνηση μιας ε, προτάσεως. Η φαιά ζώνη που αναφέρατε και επί, επ' αυτού είπε και η κυρία Κλάς κάτι για την ενημέρωση των ασθενών. Υπάρχει πράγματι αυτή η φαιά ζώνη. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα την ημέρα που υπέβαλα την δέσμη αυτή μέτρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη μεγαλύτερη ημερήσια εφημερίδα στη Γερμανία υπήρχε μια ολόκληρη σελίδα με μια συνέντευξη ενός καθηγητού ιατρικής σχετικά με ένα συγκεκριμένο εμβόλιο για την αντιμετώπιση ενός σπάνιου καρκίνου που ε, πλήγει μόνο ε, τις γυναίκες του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και το ερώτημα ήταν αν πρέπει να εμβολιάζονται τα νεαρά κορίτσια ή όχι. Με ιδιαίτερα επίμονο τρόπο συνέστησε αυτός ο καθηγητής ιατρικής την χρήση αυτού του εμβολίου. Εγώ δεν θέτω καν το ερώτημα σε ποια σχέση βρίσκεται ο καθηγητής αυτός ιατρικής με τον παραγωγό του φαρμάκου. Όμως το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε υπό την ευθύνη της αρχισυνταξίας της εφημερίδας αυτής. Εντελώς εκτός νομοθετικών πλαισίων δικών μας. Πράγματα τα οποία αποφασίζει ο αρχισυντάξης της εφημερίδας με δική του ευθύνη είναι εντελώς εκτός δικού μας ελέγχου. Και το γνωρίζετε όλοι ότι σε όλες τις δημοσιεύσεις υπάρχουν τέσσερις τομείς σε κάθε εφημερίδα, σε κάθε περιοδικό. Υπάρχουν τέσσερις τομείς όπου ποτέ δεν μπορείτε να γνωρίζετε πού βρίσκονται τα όρια μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης στο ταξίδι, στο αυτοκίνητο, στην ιατρική και στο lifestyle. Σε αυτούς τους τέσσερις τομείς, ε, δημοσιογραφικούς τομείς, ποτέ δεν μπορείτε να γνωρίζετε τι είναι τι. Γι' αυτό και μίλησα εγώ με τους φορείς και είπα ότι σε ό,τι αφορά τις πρακτικές αυτές επιθυμώ να ισχύσει ένας κώδικας δεοντολογίας και να προβλέπει αυστηρά ποια πράγματα μπορούν να γίνονται και ποια όχι. Σε αυτά πρέπει να συμμετάσχουν όμως και οι εκδότες. Δεν είναι απαραίτητα οι κακοί στην φαρμακευτική βιομηχανία, Μπορεί η κακοί να είναι και αλλού. Για το περίφημο product placement. Μπορούμε να πούμε, έχουμε, δεν έχουμε και αντίρρηση, όπω είπε ο κ. Μπόη, να μην γίνεται το product placement αυτή η έμεση διαφήμιση. Όμω αυτή η θεαζόνη, που έχει κάποια σχέση και με δεοντολογικές προδιαγραφές και στους δύο κλάδους, δηλαδή και στην ε, βιομηχανία, στον κλάδο δηλαδή των μέσων ενημέρωσης, αλλά και στον κλάδο της ε, φαρμακευτικής βιομηχανίας. Εγώ ελπίζω, και μόνο ελπίζω μπορώ, ότι ε, σήμερα όλες οι δημοσιεύσεις που υποτίθεται ότι έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα ειδικού τύπου, όπως για παράδειγμα αυτό το περιοδικό των ε, φαρμακοποιών στη Γερμανία, που εκδίδεται σε πολλά εκατομμύρια αντίτυπα και διατίθεται δωρεάν σε όλα τα φαρμακεία. Ελπίζω ότι όσα περιλαμβάνονται σε αυτό το έντυπο φροντίζει να τηρεί τα όρια τα οποία διέγραψα προλίγου. Είμαι βέβαιος και γνωρίζω καλά ότι υπάρχει αυτή η θεία Λοιπόν, λέω λοιπόν καθαρές γραμμές, ξεκάθαρα όρια και κώδικας διοντολογίας. Κύριε Ροτ Μπέρεντ, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. και για την ε, απόδοσή μου. Βέβαια όλοι μαθαίνουμε από τις προκλήσεις και ε, ε, η απόδοσή μας αυξάνεται ανάλογα με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις στην Ευρώπη. Και γι' αυτό και πρέπει να είμαστε και ε, ικανοί και αποδοτικοί. 80% των ενεργών συστατικών μέσα στα φάρμακά μας δεν παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 80%. 80% είναι εισαγόμενα. Και γι' αυτό η πρότασή μας περιλαμβάνει και διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο. Ε, εδώ όμως φέρει την κρίσιμη ευθύνη ο παρασκευαστής, ο, ο παραγωγός, ο οποίος πρέπει να φροντίσει ώστε τα ενεργα... αυτά συστατικά να μην είναι νοθευμένα και πλαστά. Ε, εν προκειμένου είμαι απολύτως ανοιχτός εάν ε, υπάρξει κάποια καλύτερη πρόταση από αυτήν που κάναμε εμείς. Για τα νάνο υλικά νομίζω ότι κατανοήσαμε η μεν τους δε. Άλλωστε θα τα πούμε και στο Στρασβούργο και θα το ξα... ξανασυζητήσουμε το θέμα. Πάντως, τουλάχιστον σήμερα, έχω την πεποίθηση ότι θα καταλήξουμε σύντομα σε μια κοινή, κοινά αποδεικτή ρύθμιση. Για τα όσα είπε και ο Αδάμου, σωστά είναι, με βρίσκουν σύμφωνο. Μια επισήμανση θα κάνω. Μου έχουν μιλήσει κατ' επανάληψη σχετικά με τα λεγόμενα φαρμακεία του ίντερνετ. Για αυτά τα φαρμακεία του ίντερνετ ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι κανόνες όπως για το φαρμακείο εδώ της γωνίας. Ακριβώς, ακριβώς οι ίδιοι κανόνες. Και λοιπόν στο φαρμακείο του διαδίκτυου πρέπει να υποβάλλεται η συνταγή εφόσον πρόκειται για, φαρμακείο, ε, για, συγγνώμη, για φάρμακο το οποίο χορηγείται μόνο κατόπιν συνταγής γιατρού, πρέπει επικεφαλής του φαρμακείου να είναι διπλωματούχος φαρμακοποιός και το καθεξής. Εάν υποπτευόμαστε, αν εσείς υποπτεύεστε ότι πρόκειται για παράθυρο μέσω από το οποίο μπαίνουν νοθευμένα φάρμακα, αυτό είναι βέβαια τότε ζήτημα ελέγχου. Όλοι βέβαια είμαστε ρεαλιστές, γνωρίζουμε ποιες είναι οι πραγματικότητες τη ζωής, γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι ορισμένα ε, φάρμακα εντός εισαγωγικών λεγόμενα lifestyle, τα οποία μάλιστα είναι ιδιαίτερα ακριβά και ε, μάλιστα ε, κανονικά χορηγούνται με σύνταγη ιατρού, περνούν από το ίντερνετ και τα παραλαμβάνει καταναλωτής χωρίς να έχει συνταγή. Βεβαίως χρειάζεται εποπτεία και έλεγχος Εάν υπάρχει εδώ νομοθετικό κενό, όσον αφορά ε, το ενδεχόμενο ανοίγματο ενός παράθυρου, όπως είπα, για την ε, εμπορία νοθευμένων φαρμάκων, ε, πάλι επαναλαμβάνω δεν είναι θέμα νομοθεσίας όσο ελέγχου της εφαρμογής της. Για την κυρία Κλάση ήδη απάντησα εν μέρη. Αυτό με το άπειρον Βεβαίω ήταν παραδρομή. Εννοούσα ότι είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και άλλωστε περί αυτού επρόκειτο στη συζήτηση ότι δεν ήθελα να έχουμε έναν απροσμέτρητο αριθμό προϊόντων, αλλά να μπορέσουμε να ρίξουμε το βάρος μας σε εκείνα των οποίων η σωστή χρήση και η ορθή παραγωγή βελτιώνουν και την κατανάλωση και χρήση ενέργειας. Έχουμε δηλαδή ήδη ενισχύει μια ρύθμιση για προϊόντα τα οποία καταναλώνουν άμεσα ενέργεια όπως ηλεκτρικές και οικιακές συσκευές και τώρα επεκτείνουμε την ρύθμιση αυτή και σε προϊόντα ή συσκευές αν θέλετε των οποίων οι χρήση έχει έμεσα πλέον κάποια επίπτωση στην κατανάλωση ενέργειας. Μόνο τέτοια προϊόντα είχε γίνει και συζήτηση αν θα έπρεπε να καταθέσουμε μια πρόταση τώρα η οποία να υπερβαίνει και τα όρια της απλής βελτίωσης της κατανάλωσης ενέργειας αλλά και να λαμβάνει υπόψη και μια προσπάθεια διατήρησης των φυσικών πόρων. Εγώ νομίζω ότι πρέπει πρώτα να συλλέξουμε εμπειρίες ε, με την εφαρμογή των προτάσεων της Κομισιόν πριν κάνουμε το επόμενο βήμα. Άρα μην ανησυχείτε το πεδίο που θέλουμε να επεκταθούμε δεν είναι άπειρο. Αυτό το άπειρο ήταν μια υπερβολή όπως συχνά μας ξεφεύγει και την κάνουμε εμείς η πολιτική. Μάλιστα, ο Πρόεδρος. Δεύτερος γύρος. Πίτερ Λίζε. Σας ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ και Επίτροπε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της ενημέρωσης και διαφήμισης για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με συνταγή. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Η φαιά ζώνη στην οποία αναφέρθηκα ο κ. Μπόης και η κυρία Κλάς δεν αναφέρεται μόνο στο θέμα της ε, ε σύναξης ε, άρθρων για καυσδημοσχεύσεις. Αλλά και μέσα στο διαδίκτυο ή μέσα στην πρόταση της Κομισιόν υπάρχουν φαίες ζώνες. Και η Κομισιόν λέει ότι οι πληροφορίες οι οποίες είναι δυνατόν να χορηγούνται κατόπιν της πρότασης δεν είναι θέμα διαφήμισης. Αλλά είμαστε σε διαδικασία συναπόφασης και υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι που λέμε ότι ένα τμήμα των πληροφοριών που θέλει να χορηγήσει ελεύθερα η Κομισιόν θα μπορούσαν να θεωρηθούν διαφήμιση. Και στην συναπόφαση το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι αυτό το σημείο να το διευκρινίσουμε, να το περιορίσουμε ώστε ε, με καθαρή συνείδηση να μπορούμε ότι δεν πρόκειται για, α, για άρση της απογόρευσης διαφήμισης, αλλά πρόκειται για ενημέρωση. Αλλά είδαμε πάντως κάθαρα ότι και στο ιστορικό της Κομισιόν μία επίτροπος που είναι αρμόδια για θέματα ε, υγείας έχει υποβάλει πολύ πιο συγκεκριμένε προτάσεις. Λοιπόν, άλλο θέμα εδώ σχετικά και στην περασμένη θητεία όταν είχαμε μια παρόμοια πρόταση είχα πει ότι εκπρόσωποι των ασθενών θα πρέπει στην ε, νομοθεσία να θεωρηθούν ισότιμα με τους γιατρούς. Γιατί πραγματικά εκπρόσωποι των οργανώσεων αυτών αυτοβοήθειας των ασθενών είναι πολύ πιο ενημέροι από, ένας μέσο, από ένα μέσο γιατρό, ιδίως στο θέμα των σπανίων ασθενειών. Αλλά θα πρέπει να δούμε όταν εδώ ασθενείς ή οργανώσεις αυτοβοήθειας των ασθενών θεωρούνται γιατροί και δίνουμε περισσότερες πληροφορίες από εκείνους που δίνουμε στο ευρύ κοινό. Πώς θα αποφύγουμε εκείνες οι οργανώσεις άλοθη γιατί ορισμένες ε, λειτουργούν σαν μέσο της φαρμακοβιομηχανίας. Πώς θα κάνουμε λέω τη διάκριση γιατί είναι πολύ δυσάρεστο η Κομισιόν να καλεί αυτού τις οργανώσεις αλλά σε ακροάσεις και άλλες οργανώσεις να μην μπορούν να τοποθεθούν. Πώς θα μπορούμε αυτές οι οργανώσεις των ε, ασθενών να ε, έχουν μια εξάρτητη χρηματοδότηση και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τελευταίο σημείο. Δικαίως αναφερθήκατε στο ότι θα πρέπει πάντα να αιτιολογεί κανένας γιατί δεν δίνει κάποιες πληροφορίες. Και εδώ αναφέρομαι στα was so normalerweise im Beipackzettel steht, nicht einfach zu verstehen Στις οδηγίες χρήσεως που υπάρχουν μέσα στα φάρμακα υπάρχει και η δυνατότητα των οδηγιών αυτών συν. Και άμα πούμε τώρα γιατί δεν θέλουμε γενικά να το έχουμε αυτό όταν λέμε δηλαδή ότι είναι θέμα της βιομηχανίας ε, του κλάδου ελεύθερα να δίνει συμπληρωματικές πληροφορίες οδηγίες αυτές, γιατί δεν μπορούμε να το πούμε ξεκάθαρα, ότι να πρέπει να δίνεται ένα φάρμακο μόνο με μία εύκολα κανατοητό συνοδευτικό έγγραφο, ευνόητο, εύληπτο και όχι αυτά τα χαρτιά που υπάρχουν σήμερα, γιατί αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τον ασθενή. Θα θέλω να πω την άποψή σας από αυτού. Thank you very much indeed. Uh, σας ευχαριστώ. Η Λίντα Μακάβαν. Ευχαριστώ. Πριν σχολιάσω τι παρατηρήσει του κ. Μπόση και τι δικέ κ. Επιτροπή για τα φαρμακευτικά προϊόντα και το έργο που επιτελεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την πράσινη, το πράσινο πρόγραμμα εργασιών τη, νομίζω ότι πολλά κάνει και ίσω κάπου θα πρέπει να συντονιστούν οι διάφορε υπηρεσίε για να μπορέσει ο πολίτη να έχει μια συνολική εντύπωση για το τι κάνει η Επιτροπή και οι διάφοροι Επιτροπηδοί μας μακρύβοι εσείς. Θα πρέπει να συνδυάσουμε ώστε να μπορέσει και ο να αντιληφθεί ε, το παράλληλο έργο μερικές φορές διαφορά γενικών διευθύνσεων. Είναι πολύ σημαντική αυτή η νομοθετική πρόταση και νομίζω ότι εκεί πραγματικά μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να περιορίσει τις ενεργειακές δαπάνες και να μειώσει το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Είναι πολύ σημαντικές οι προτάσεις που κάνατε για την ενεργειακή εξοικονόμηση. Ό,τι αφορά την ε, εποπτεία, επιτήρηση για τα φάρμακα, επαγρύπνηση για τα φάρμακα, είναι πολύ σημαντικό και αυτό το θέμα. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, γιατί δεν θα προλάβουμε στην κοινοβουλευτική μας θητεία να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Θα το αναλάβει το επόμενο κοινοβούλιο. Τώρα, εγώ είμαι ένας κοινό άνθρωπος. Ε, λέτε ότι θέλετε δίπλα στα φάρμακα να, έχει, να υπάρχει και ένα ειδικό ενημερωτικό ε, τμήμα για τις παρενέργειες. Ποιος είναι αυτός ο στόχος ε, της αλλαγής για έναν κοινό άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει. Γιατί φαίνεται ότι η φαρμακευτική βιομηχανία είναι μάλλον κατά της ιδέας. Και ένας απλός πολίτης θα μπερδευτεί. Γιατί Αναφέρονται όλες οι παρενέργειες, οπότε βλέπουμε έναν ε, τεράστιο κατάλογο, μακροσκελέσταλο κατάλογο ε, παρενεργειών, αλλά δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει ένα ποσοστό πιθανότητων για κάθε παρενέργεια. Οπότε αυτό έχει το αντίθετο αποτέλεσμα μερικές φορές. Και εγώ είχα μια πολύ αρνητική αντίδραση και νομίζω ότι 30% των ε, ανθρώπων που αγοράζουν τα φάρμακα διαβάζοντας αυτόν τον ε, εκτενέστατο κατάλογο των παρενεργειών την ίδια αντίθετη αντίδραση έχουν. Τελικά βλέποντας όλο αυτό το κατάλογο δεν προσέχουν καθόλου τις παρενέργειες και αισθάνονται πολύ πιο μπερδεμένοι οι απλοί πολίτες. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το εξετάσετε για να αποφύγουμε αυτό το dumping της πληροφόρησης, να γίνει σωστή ενημέρωση, αλλά να αποφευθεί αυτό το dumping που ήδη ισχύει. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο. Και πάλι για την ενημέρωση του ε, ασθενούς είχαμε με τον κύριο Φιέλνερ, ε, τον εισηγητή μας, εκτενή ζήτηση την περασμένη εβδομάδα. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει ένα τρίτο αμερόληπτο, αμερόληπτο ε, μέρος που να δίνει αυτές τις πληροφορίες για τα φάρμακα και όχι οι ε, συγκεκριμένες φαρμακοβιομηχανίες. Προτάθηκε λοιπόν αυτή η ιδέα ένα τρίτο ανεξάρτητο να δίνει αντικειμενικέ αμερόληπτε πληροφορίε για τα φάρμακα σε ένα επιστημονικό περιοδικό, για παράδειγμα, και τι διάφορε ε, συνθήκε των θεραπείων. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα βοηθήσει να έχουμε ένα τρίτο ανεξάρτητο μέρο που να, δίνει αυτές τις, να παρέχει αυτέ τι αντικειμενικέ πληροφορίε για να επιλύσουμε και το θέμα τη ε, φεαζόνη. Ο κύριο Κράμερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ γλυγορά. Έχω δύο ερωτήσει όσον αφορά τα φάρμακα. Θα αρχίσω με την ενημέρωση των ασθενών. Το είπα και την περασμένη εβδομάδα. Γενικά έχω την εντύπωση ότι η πρόταση τη Κομισιόν θα μα βοηθήσει να προχωρήσουμε γιατί ε, αλαφρύνει μια απόλυτη απογόρευση πληροφορία που, που ισχύει αυτή τη στιγμή και την διαχωρίζει και από την απογόρευση της διαφήμισης. Δεν πρέπει όμως να έχουμε τις ψευδεθήσεις ότι θα μπορούσαμε να εξαλείψουμε όλες τις φαιές που υπάρχουν μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τα πάντα. Κάποιες σφαίρες ζώνες θα παραμείνουν. Και θα πρέπει βέβαια να φροντίσουμε στο τέλος να μην έχουμε τόσο στενούς περισμούς που να μην έχουμε καμία ενημέρωση. Πάνω στην πρόταση Κομισιόν έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. η πρόταση προβλέπει απαγόρευση σύγκρισης μεταξύ φαρμάκων. Είναι λογικό αυτό. Να μην επιτρέπεται να υπάρχει σύγκριση μεταξύ φαρμάκων, γιατί οι ασθενεί συνήθω δεν έχουν τι γνώσει για να μπορούν να αξιολογήσουν τη σύγκριση αυτή. Αλλά η πρόταση αφήνει ανοιχτό ένα παραθυράκι. Δηλαδή, συγκρίσει μεταξύ φαρμάκων είναι δυνατές εάν δοθούν στο γιατρό και ο γιατρός τους δώσει μετά στον ασθενή. Κατά πόσο είναι κάτι τέτοιο λογικό. Γιατί έτσι ο ασθενής δεν έχει καμία δυνατότητα να εξετάσει και άλλα συγκριτικά στοιχεία. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εκεί. Δεύτερο θέμα και συμφωνώ. Απόλυτα εδώ με την κυρία Ροτ Μπέρεντ ότι συζητάμε εδώ πλαστά φάρμακα και όχι παράνομο εμπόριο. Α, συμφωνώ απόλυτα. Θα πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα μέτρα που θα εθοδίσουμε εδώ να στοχεύουν συγκεκριμένα στα πλαστά φάρμακα χωρίς να πλήξουν ταυτόχρονα και ένα παράλληλο εμπόριο. Πάνω σε αυτό νομίζω συμφωνούμε γιατί εδώ, το λέω αυτό, αριστερά πίσω από μένα, υπάρχουν πολλοί εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας που καμιά φορά θέλουν ας πούμε, να χρησιμοποιήσουν αυτού του είδους την νομοθεσία για να απαγορεύσουν μία οδό εμπορίας που δεν τους είναι πάρα πολύ προσφύλης. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί που βρίσκεται το επίκεντρο της συζήτησης μας. Και σας θέλω να ρωτήσω το εξή ότι η Διεθνής Οργάνωση Υγείας ε, δημοσίευσε αποτελέσμα το 50% των πλαστών φαρμάκων που ε, βρίσκονται στο εμπόριο περνάνε μέσα από το διαδίκτυο, από το ίντερνετ. Πιστεύετε η νομοθεσία που προτείνεται θα αρκήσει αρκέσει για να περιορίσει πραγματικά, για να απογορεύσει αυτό το εμπόριο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κουτιέρες Κορτίνες θα είναι τελευταία τελευταία ομιλήτρια του δεύτερου γύρου των ερωταπαντήσεων. Έχετε το λόγο κυρία Γκουτιέρες. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερο και συγχαίρω τον Επίτροπο, γιατί πριν από ένα-δύο χρόνια η κυρία Σαρδόρη και εγώ εκπονήσαμε ένα ψήφισμα για τις ε, δραστικές ουσίες ε, εισαγωγής και την έλλειψη ελέγχου και χαίρομαι που στην τελευταία της πρώτης Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέλαβε και τον έλεγχο της εισαγωγής των ενεργών δραστικών ουσιών των φαρμάκων. Μπράβο σας κύριε Επίτροπε, σας μεταφέρω και τα συγχαρητήρια της κυρίας Αρτόρη που απουσιάζει σήμερα. Δύο όμως ε, ανησυχίες έχω για το θέμα αυτό. Παρόλο που είναι προφανές ότι με ένα-δύο έγγραφα δεν πρόκειται να επιλύσουμε όλα, όλες τις τρευλώσεις της αγοράς. Ερωτώ λοιπόν, πώς θα αποφύγουμε το πρόβλημα που έχουμε με τη σύγκρουση την αναποτελεσματικότητα της διανομής των φαρμάκων. Γιατί μερικές φορές για κάποια συμφέροντα, λόγω της αναποτελεσματικής οργάνωσης αγοράς, έχουμε, όπως συνέβη φέτος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, έλλειψη φαρμάκων, σπάνι φαρμάκων. Τέτοιο φαινόμενο παρατηρήθηκε φέτος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια στιγμή κυρία Κουτιέρες Κορτίνες. Παρακαλώ λίγη ησυχία, μη συνομιλείτε εντός της γιατί γίνεται μεγάλη φασαρία και δεν μπορούμε να ακούσουμε. Συνεχίστε κυρία Κουτιέρες Κορτίνες. Δεύτερο θέμα. Εσείς κύριε Επιτροπή, αλλά και άλλη Επιτροπή, ταχθήκατε υπέρ της απελευθέρωσης των φαρμακείων. Ενώ είναι σαφές ότι ο φαρμακοποιός είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ε, δώσει συμβουλές στους ηλικιωμένους και να ενημερώσει έναν ασθενή για συμβατότητες μεταξύ διαφόρων φαρμάκων που πολλούνται μερικές φορές και χωρίς ιδέα όπως η ασπιρίνη. Ασπιρίνη όμως δεν μπορεί να πάρει κάποιος καρδιοπαθής που έχει ε, υποστεί και επέμβαση καρδιάς. Γιατί λοιπόν να απελευθερωθούν τα φαρμακεία. Γιατί ο φαρμακοποιός είναι αυτός που θα δώσει πληροφορίες. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει το ίντερνετ. Δεν μπορεί να έχει άμεση επαφή ο φαρμακοποιός μέσω ίντερνετ και να συμβουλέψει πραγματικά τον ασθενή. Ευχαριστώ. Äh, äh, äh, Ο Επίτροπος. Κύριε Λίζε, ευχαριστώ για τη διευκρίνηση σχετικά με το τι εννοούσατε. Μου φαίνεται κάπως φιλικότερο τώρα αυτό που είπατε από αυτά που διάβασα αρχικά από εσά. και μπορώ να συμφωνήσω και περισσότερο. Αν θέλετε να μου πείτε ποιες είναι οι οργανώσεις εκείνες ασθενών που δεν είναι τίποτε άλλο παρά κατά κάποιο τρόπο ε, παρατρεχάμενοι των φαρμακευτικών βιομηχανιών, ε, θα δω πώς θα αντιδράσω και θα αντιδράσω σίγουρα. Σε ό,τι αφορά τις οδηγίες των φαρμάκων, θεωρώ ότι οι πληροφορίες που παρέχει ο ε, παραγωγός του φαρμάκου και που πρέπει να είναι εγκεκριμένο βεβαίως δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά αυτά που θέλει να προσφέρει με ένα ευανάγνωστο τρόπο ως υποπροϊόν της ε, πρότασής μας θα είναι και αυτό Μάλιστα πρόσφατα χρησιμοποίησα ένα φάρμακο, διάβασα το ε, χαρτάκι και ήταν πραγματικά κατανοητό ήταν μάλιστα συνταγμένο σε ορότατα γερμανικά και διερωτήθηκα γιατί δεν τα κάνουμε όλα έτσι. Ε, διότι έχει σχέση με θέματα ευθύνη, όπου για να είναι καλυμμένοι σε κάθε περίπτωση ευθύνη χώνουν τα πάντα μέσα. Έχω λοιπόν μεγάλη κατανόηση ε, σχετικά με την πρόταση να βελτιωθεί η ποιότητα. Αυτό πρέπει να συζητηθεί βέβαια και με την αρχή έγκρισης των φαρμάκων. Κυρία Μακάβαν, θα φροντίσω ώστε να λάβετε δέσμη πληροφοριών σχετικά με το Green Procurement, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και ε, τι μπορούμε να κάνουμε ακόμη. Θα σας τα διαβιβάσουμε ήδη μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά την εποπτεία για τη χρήση των φαρμάκων, δεν πρόκειται για κινδύνους μόνο γνωστούς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την επιτήρηση, την εποπτεία των φαρμάκων είναι να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να μας πληροφορεί, να μας ε, ενημερώνει, να κρούει ένα κόδωνα όταν εμφανίζονται κίνδυνοι που δεν γνωρίζουμε. Ε, αναλόγως του αν είναι κεκριμένο το φάρμακο, αν χορηγείται μόνο με συνταγή ιατρού ή όχι, και άλλα στοιχεία που μπορεί να είναι χρήσιμα για την χρήση ενός φαρμάκου και βεβαίως διασυνδέονται με τους κινδύνους. Πολλά φάρμακα, τα οποία μάλιστα έχουν και επικίνδυνες παρενέργειες, ορισμένα εξ αυτών, και επομένως δεν μπορούν παρά να χορηγούνται σε πολύ ειδικέ περιπτώσεις οι σχετικές πληροφορίες είναι βεβαίως γνωστές σε όλους τους αρμόδιους. Μιλώ όμως για κινδύνους που δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα μπορεί να αποδειχτεί και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και τραγικές περιπτώσεις όπου συνέβησαν τέτοια πράγματα, όπου δηλαδή εμφανίστηκαν κίνδυνοι ή κατέστησαν γνωστοί κίνδυνοι όταν το φάρμακο ήδη ήταν σε κυκλοφορία και χρησιμοποιήθηκε για ορισμένες, για, κάποιο χρονικό διάστημα. Μιλούμε λοιπόν για νέους νεοαναφαινόμενους κινδύνους ή ε, ενδεχομένως που προκύπτουν σε συνδυασμό με κάποιον άλλο κίνδυνο. Είναι χρήσιμο αυτή η πληροφορία να φτάνει με ταχύτητα στις αρμόδιες αρχές ώστε να μπορούν αυτές να αντιδρούν λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα. Για την δυνατότητα να παρεμβαίνει και ένα ανεξάρτητο πρόσωπο στην ενημέρωση του ε, ασθενούς. Θα το κοιτάξουμε, αλλά το δικαίωμα το οποίο παραχωρείται στους παραγωγούς φαρμάκων να ε, διοχετεύουν πληροφορίες μέσω των δημοσιεύσεων σε περιοδικά κτλ. Έχει βεβαίως και σχέση με το ότι αυτοί κάτι πληρώνουν για να δημοσιευτεί το σχετικό άρθρο. Όταν θέλω ως μεγάλος παραγωγός φαρμάκου να δημοσιεύσω κάτι σε ένα μεγάλο επιστημονικό περιοδικό, τότε υπάρχουν δύο δυνατότητες. Είτε γίνεται υπό την ευθύνη της αρχισυνταξίας, οπότε εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε, είτε εμφανίζεται υπό την ευθύνη του παραγωγού. Και αυτό βεβαίως πρέπει αφενός να επισημαίνεται στο άρθρο, και αφετέρου ελέγχεται ο παραγωγός. Βεβαίως δεν είναι δωρεάν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω λοιπόν πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα σύστημα όπου θα παρεμβαίνει και ένα τρίτο ουδέτερο πρόσωπο. Μιλούμε εν προκειμένου δηλαδή για εκ των προτέρων έλεγχο των πληροφοριών. Δηλαδή πρέπει να εγκριθεί πρώτα η πληροφορία πριν να δημοσιευτεί. Κύριε Κράμερ, ομολογώ ότι δεν μπορώ να απαντήσω στην πρώτη σας ερώτηση. Άλλωστε δεν έχω και το κείμενο μπροστά μου. Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω γραπτός λοιπόν εν ε, προκειμένου αν χρειάζεται διευκρίνηση στο κείμενο βεβαίως ε, τα κείμενά μας δεν θεωρώ ότι είναι απολύτως αλάθητα μιλήσατε και, και εσείς για το εμπόριο μέσω ίντερνετ. Εάν βεβαίω, βεβαίως κάποιος είναι ανόητος, ένας Ευρωπαίος καταναλωτής είναι τόσο ανόητος ώστε να αγοράσει, να παραγγείλει ένα φάρμακο μέσω του ίντερνετ στην Ιγυρία, ε τότε τι να κάνω κι εγώ, πώς να τον βοηθήσω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθήσω να ενημερώσω τον κόσμο, προσέξτε, μην παραγγέλνετε τα φάρμακά σας ε, από προμηθευτές εκτός ευρωπαϊκών χωρών και κυρίως από χώρες όπου γνωρίζουμε ότι το 50% των φαρμάκων ούτως ή άλλως είναι αθευμένα. Έχουμε εδώ την ίδια περίπτωση όπως και με το παράλληλο εμπόριο. Στο παράλληλο εμπόριο μπορεί κανείς να έχει βέβαια διαφορετικές Αντιλήψει σχετικά με την οικονομική ωφέλεια του παραλληλού εμπορίου, μπορεί κανείς εκεί να διαφωνεί εν πάση περιπτώσει. Αλλά ε, όταν από τη σκοπιά μια μεγάλη χώρα μέρους όπως η Γερμανία, το παράλληλο εμπόριο είναι μια ε, χρήσιμη δραστηριότητα και καλοδεχόμενη, διότι μειώνει το κόστος της υγείας. Από τη σκοπιά της Πορτογαλίας, για παράδειγμα, το παράλληλο εμπόριο δεν είναι απαραίτητα χρήσιμη δραστηριότητα, διότι οδηγεί ώστε στην Πορτογαλία να μην είναι διαθέσιμα ορισμένα φάρμακα. Πώς να σταθμίσει κανείς τι γίνεται σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο εγώ δεν έχω πλέον τη δυνατότητα καν να προβώ στη στάθμιση αυτή διότι η απόφαση του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι σαφής. Λέει ότι υπερέχουν οι κανόνες της ενιαίας αγοράς ακόμα και σε φάρμακα τα οποία χορηγούνται μόνο με συνταγή ιατρού. Εφόσον η απόφαση του δικαστηρίου δεν πείται διάκριση ανάμεσα σε φάρμακα τα οποία χορηγούνται με ε, ιατρική συνταγή και σε παιδικά ποδήλατα. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να τηρήσουμε το ισχύον δίκαιο. Και εν προκειμένου το ίδιο. Έχουμε λοιπόν μονοσήμαντη νομολογία, δεν μπορούμε να περιορίσουμε το ε, εμπόριο μέσω διαδικτύου, ούτε και για φάρμακα. Παρόλο που εγώ ο ίδιος έχω μεγάλες αμφιβολίες εάν είναι πραγματικά απολύτως δυνατό να ελέγχεται το φαρμακείο του ίντερνετ. Τον έλεγχο βεβαίως αναλαμβάνουν να κάνουν οι μέλη. Πρέπει να ελέγξουμε και πάλι ε, πώς έχει το θέμα και να επανέλθουμε. Εάν ορισμένες ε, μορφές προμήθειας για φάρμακα με συνταγή γιατρού. Μήπως θα έπρεπε να υπακούν, να υποτάσσονται σε κάποια άλλη προτεραιότητα και όχι απαραίτητα στην υπεροχή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες εν προκειμένου. Εάν δηλαδή πρέπει εν πάση περιπτώσει η ελευθερία διακίνησης των εμπορευμάτων μέσα στην ενιαία αγορά να είναι απόλυτα η πρώτη απόλυτη προτεραιότητα ή μήπως υπάρχουν κάποια αντικείμενα τα οποία ε, στην περίπτωση των οποίων δηλαδή θα πρέπει για παράδειγμα ε, κανόνες ασφάλειας να έχουν ένα ε, σημαντικότερο ρόλο, πλεονεκτικότερο ρόλο. Πρέπει άλλωστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την εισρωή και πλαστών υνοθευμένων φαρμάκων από τρίτες χώρες με έλεγχο να υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες αλλά είμαι διατεθειμένος να διαβουλευθώ περαιτέρω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θεωρώ ότι έχει κεντρική σημασία. Για να μην παρεξηγηθούμε, η πρόταση που έχουμε κάνει αναφέρεται στην ασφάλεια κατά ε, πλαστών υνοθερμιών φαρμάκων μέσα στη νόμιμη διακίνηση του φαρμάκου. Δεν έχει νόημα να επαναλάβουμε την απαγόρευση ε, νοθείας κτλ. Μιλούμε τώρα για ε, τη νόμιμη εμπορία του φαρμάκου, για την παράνομη εμπορία. Αυτό είναι θέμα βέβαια εφαρμογής του δικαίου και καταπολέμησης του εγκλήματος. Για σας κύριε Γκουτιέρες, είναι όντως δυσχερές θέμα και δεν μπορώ να το συζητήσω αφηρημένα. Κατ' επανάληψη, ε, συμβαίνει σε ορισμένες αγορές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κάποια φάρμακα να μην είναι διαθέσιμα. Ε, και είναι ένα ε, πρόβλημα το οποίο επανέρχεται για παράδειγμα σε πολύ μικρές αγορές όπως Μάλτας και Κύπρου λόγω και του ορισμού να ε, περιλαμβάνεται το φυλάδιο ε, με τις οδηγίες και στην τοπική γλώσσα της χώρας δηλαδή, όπου για ορισμένους ε, παραγωγούς δεν έχει ενδιαφέρον οικονομικό, επειδή είναι τόσο μικρή αγορά. Και όμως λόγω της δράσης του παράλληλου εμπορίου είναι δυνατόν να μην είναι διαθέσιμο ένα φάρμακο διότι ε, για παράδειγμα οι αρμόδιες ε, αρχές της ε, χώρας εκείνης δεν το έχουν περιλάβει μεταξύ, στον κατάλογο των φαρμάκων εκείνων τα οποία, για τα οποία επιστρέφονται οι δαπάνες. Μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα βέβαια. Η πρότασή μας δεν έχει βέβαια σχέση, καμία σχέση με απελευθέρωση ε, της αγοράς των φαρμάκων. Βλέπω ότι μπορεί εδώ να ελευθερωθεί εν προκειμένου. Δεν ξέρω πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχει κάποια παρανόηση. Ασφαλώς και παραμένουν ενισχύει οι αυστηρές προδιαγραφές για την θέση κυκλοφορία των φαρμάκων, ε, οι διατάξεις σχετικές με την ευθύνη και ούτω καθεξής. Δεν ε, βλέπω που ίσως ε, θεωρείτε ότι παρισέφθησε κάποιο στοιχείο απελευθέρωσης της αγοράς. Εγώ δεν βλέπω τίποτα τέτοιο. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Πριν τον τελευταίο γύρο των ομιλητών, να σας ε, ανακοινώσω ότι έχουμε ξεπεράσει το ωράριό μας. Βέβαια το περίμενα. Γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω να είστε όσο πιο λακωνικοί γίνεται. Ο Τόμας Όρμαρ πρώτα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα είμαι σύνομος για την επιτήρηση των φαρμάκων. Δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα, αλλά θα ήθελα να μην είναι ένα κράτος μέλος που εκείνο που δηλώνει κατά 95% τις περιπτώσεις και άλλους κόσμος να μην δηλώνει τίποτα. Τα ξέρουμε αυτό και άλλους ε, τομείς. Όσον αφορά τα πλαστά φάρμακα, επίσης δεν βλέπω να υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι για τις παράλληλες εισαγωγές να βρούμε μια καθαρή λύση. Και ε, βλέπω ότι θα ήταν καλό πραγματικά εδώ να ε, υπάρχει πιο ενωπημένη αγορά, ιδίως και προς όφελος των ε, καταναλωτών, των ασθενών, που μπορούν παντού να βρίσκουν τα φάρμακά τους θα μπορεί να υπάρχει σχετική οργάνωση των κρατών μελών, αλλά δεν είναι θέμα αρμοδιότητας μας. Όσον αφορά την ενημέρωση των ασθενών, προφανώς όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν όλες τις πληροφορίες στα χέρια τους. Το περιγράψα μας πάρα πολύ ωραίο ότι καταφέρετε να καταλάβετε ένα από τα συνοδευτικά αυτά χαρτάκια επειδή ήταν καλά και σαφώς διατυπωμένο γιατί πραγματικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το θέμα της ε, πληροφόρησης είναι αυτό που φτάνει στον καταναλωτή και όχι εκείνο που αποστέλλεται από τον αποστολέα. Θα πρέπει να διακανονίσουμε το θέμα της ενημέρωσης ε, των ασθενών, αλλά δεν θα διακανονίσουμε εδώ το θέμα της σχέσης γιατρού και ασθενούς. Αυτό το αφήνουμε κατά μέρος. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μην επιβαρύνουμε με γραφειοκρατικά μέτρα ή κόστος συμπληρωματικό όλους τους ε, φορείς του ε, υγειονομικού τομέα. <clears throat> Όσον αφορά το θέμα της ε, διάκρισης μεταξύ διαφήμισης και ενημέρωσης, αναφέρθηκατε στο καλό αυτό παράδειγμα του περιοδικού αυτού που δίδεται στα φαρμακεία στη Γερμανία. Από την άλλη μεριά βέβαια, ε, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να παρατείνουμε τη ζωή των ε, ασθενών. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες ε, των εμβολίων για την υποτίτητα Β, παραδείγματος χάρη μετά από τη, το γεγονός ότι υπήρχαν διευρυμένες εκστατείες εμβολίων, 40.000 ασθενείς λιγότεροι πεθαίνουν το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας που θα είναι αποχρεώνει όλους τους ενδιαφερομένους και εμπλεκόμενους να αντιμετωπίσουν τα πράγματα σωστά. Θα υπάρχουν πάντα ακραίε περιπτώσει και οριακέ περιπτώσει, αλλά νομίζω ότι με το φάκελο αυτό προχωρούμε προ τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Ντόιλ είναι το λόγο. Thank you and thank you. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τον Επίτροπο που μας αφιέρωσε γενναιόδωρα το απόγευμά του. Ο Τζον Μπόις αναφέρθηκε στη θεά ζώνη μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης ή διαφήμισης και ενημέρωσης. Υπάρχει και μια άλλη θεά ζώνη που θα ήθελα να μας διαλευκάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τη σχολιάσει. Η θεά ζώνη στη συζήτηση του τι εστί φάρμακο και τι εστί φαρμακευτικό εξοπλισμός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα και συναφές με τα φαρμακευτικά προϊόντα. Γιατί η παραχώρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την πρόταση αναδιατύπωση της οδηγίας για το φαρμακευτικό εξοπλισμό οι φαρμακευτικές συσκευές. Περιμένουμε την αναδιατύπωση της σχετικής οδηγίας. Επίσης έχουμε και το κατευθυντήριο όργανο ΜΕΝΤΕΦ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ορίζει τη διαφορά μεταξύ φαρμακευτικής συσκευής και ε, ιατρικής συσκευής. Υπάρχει σημαντική νομολογία στην Γερμανία εξαιτία της διαφοράς ερμηνείας. Υπάρχει ε, διαφορά μεταξύ των εθνικών ερμηνεών αλλά και διασυνοριακά δημιουργώντας μια τεράστια σύγχυση μεταξύ του διαχωρισμού ιατρικών συσκευών και φαρμακευτικών. Πριν από 10 χρόνια είχαμε την οδηγία για τις ιατρικές συσκευές που έχει γίνει πλέον απερχιωμένη γιατί υπήρξε τεράστια τεχνολογική εξέλιξη και επιστημονική εξέλιξη γενικώ για τις ε, ιατρικές συσκευέ και τον ιατρικό εξοπλισμό. Ε, επίσης, ε, ε ένα χάπι για παράδειγμα κατά της δυσκυλιότητας θεωρείται φάρμακο ή ε, συσκευή φαρμακευτική. Θα πρέπει να επιταχύνεται τις εργασίες για την αναδετύπωση της οδηγίας ε, μεταξύ ε, τις που καλύπτει τις ιατρικές συσκευέ και τα φάρμακα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Η κυρία Κάθη Σίνοτ. Ευχαριστώ. Έχω τρεις ερωτήσεις κύριε Επίτροπε. Μιλούμε για την όλο και περισσότερο πράσινη φιλοπεριβαλλοντική πτυχή της οικονομίας. Γιατί είναι δύσκολο να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος της φιλοπεριβαλλοντικής οικονομίας. Και στην πατρίδα μου έχω συναντήσει και έχω συνεργαστεί με πολλούς ανθρώπους που έχουν φαϊνές ιδέες για την παραγωγή βιοκαυσίμων, για την πράσινη οικονομία και δεν μπορούν να υλοποιήσουν τους στόχους τους γιατί η εταιρεία φυσικού αερίου είναι ιδιοκτήτρια για την ε, μεταφορά φυσικού αερίου και έτσι δεν δίνει άδεια και δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να παράγουν βιοκαύσιμα. Δεν ε, εντάσσονται στο δίκτυο και έτσι όλα τα σχέδια που υποβάλλουν είναι πολύ εφάνταστα ήδη από τα σπάργανά τους αναβαγούν. Το ίδιο και στον ηλεκτρισμό. Θέλουμε να υπάρχει διαφοροποίηση στην αγορά. Μην έχουμε μόνο τις μεγάλες ε, εταιρείε παραγωγής ηλεκτρικού, γιατί έτσι η τοπική πρωτοβουλία ασφικτιά, γιατί δεν εντάσσεται στο δίκτυο των μεγάλων εταιρείων. Άλλωστε οι εταιρείε αυτές φυσικού αερίου κυρίως δουλεύουν με ε, καύσιμα, με ορυκτά καύσιμα και προσπαθούν να διονύσουν αυτή την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα χωρίς να δώσουν καμία ευκαιρία στα βιοκαύσιμα. Κάναμε τεράστιες προσπάθειες για τα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και αυτό είναι το ίμιση της ιστορίας, γιατί θα πρέπει να δαχθούμε ε, μαθήματα από αυτή την εμπειρία μας. Θα πρέπει να δώσουμε και τη διάρκεια ζωής ενός τέτοιου ενεργειακού αποδοτικού προϊόντος σε ώρες, θα πρέπει να γίνει με τέτοια ποσοτικοποίηση. Και τέτοιου είδους στοιχεία θα πρέπει να υπάρχουν στο πακέτο. Όταν ένα προϊόν είναι ενεργειοβόρο θα πρέπει να αντικαθίσταται από ένα πιο αποδοτικό ενεργειακά προϊόν. Επίσης έχω απογοητευτεί και το θέμα των ρυθμιστικών αρχών για τα φάρμακα. Μιλήσατε για την προστασία της ασφάλειας, για την αναχέτηση της ε, παραγωγής των πλαστών φαρμάκων. Εμείς όμως έχουμε ακόμη και στο ε, δίκτυο ίδρευσης ε, το δημοτικό ουσίες που κυκλοφορούν χωρίς να έχουν αδειοδοτηθεί. Έχουμε μια τέτοια ουσία που κυκλοφορεί στο πόσιμο είδωρο από τα 50, δεν έχει λάβει άδεια για να κυκλοφορήσει ως φάρμακο και παρόλο που έχει χαρακτηριστεί από την νομοθεσία ως φάρμακο η ουσία αυτή. Και οι υγειονομικές υπηρεσίες το έχουν, έχουν εισαγάγει αυτή την ουσία στο υδροδοτικό δίκτυο. Με σημαντικές παρενέργειες μακροχρόνια για τους Ιρλανδούς πολίτες. Τα έχω επισημάνει επανειλημμένο σε αυτό το σκάνδαλο τα τελευταία 4,5 χρόνια, αλλά δυστυχώ όλα μου τα σχόλια έχουν αγνοηθεί. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Βέικμαν είναι ο τελευταίος μας ομιλητής. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Έφτασα αργά στην συνεδρίαση. Μπήκα όμως στην αίθουσα την ώρα που μιλούσατε για την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό και χαίρομαι για τα σχόλιά σας. Σε αντίθεση με την Κρίστα Κλάς, δεν πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επεμβαίνει σε όλες τις ε, μεμονωμένε οδηγίες. Χρειαζόμαστε μια οδηγία πλαίσιο και να επικεντρωθούμε σε φιλο... φιλοπεριβαλλοντικά προϊόντα που έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Δεν έχουμε εδώ ενδιαφέρον μόνο για την χρήση της ενέργειας. Πριν από λίγα χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε σε ένα εγγραφό τη ότι η χρήση των φυσικών πόρων γενικά είτε είναι παραδοσιακές πηγές είτε ανανεώσιμες πηγές θα δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον και αυτό το δήλωσαν και οι επιστήμονες όχι γιατί έχουμε πολλές αναφιόμενες οικονομίες παντού στον κόσμο που αναζητούν πρώτες ύλες γιατί πολλές τέτοιες χώρες αναφιόμενες οικονομίες θέλουν να εξασφαλίσουν ε, τα ορυχεία τους, την υλοτομία τους ε, και τις πρώτες ύλες τους από την Αφρική. Βέβαια στο παρελθόν έγιναν κάποιες απόπειρες για την ενθάρρυνση της ε, επαναχρησιμοποίησης της ανακύκλωσης, αλλά ελάχιστα τελικά ήταν τα επιτεύγματά μας στον τομέα αυτό. Και η παρούσα οργάνωση της παραγωγής και της κατανάλωσης δεν είναι βιώσιμη θα πρέπει να έχουμε μια πιο λειτουργική οργάνωση. Αντί να αγοράζουμε ένα προϊόν, να το μισθώνουμε ή να το εκμισθώνουμε. Έτσι θα είχαμε πολύ διαφορετικό τοπίο. Επίσης θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο τις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφοριών ή να μιμηθούμε τη φύση χρησιμοποιώντας ε, περισσότερα απόβλητα, ανακυκλωμένα απόβλητα όλο και περισσότερο ανακυκλωμένα υλικά. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να προωθήσετε αυτό το πρόγραμμα περισσότερο. Γιατί δεν άρχισε σήμερα η συζήτηση για το θέμα αυτό, αλλά πριν από μία δεκαετία για την ολοκληρωμένη πολιτική για τα προϊόντα. Αλλά ελάχιστη ήταν η πρόοδος μας. Τώρα έχουμε μία οδηγία με πολύ καλή μεθοδολογία και θα μπορούσαμε κάλλιστα να περιλάβουμε όλα τα μέτρα για την ε, αποδοτικότητα της ενέργειας και την αποτελεσματικότητά της. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, έχετε το λόγο. Θα είμαι σχετικά σύντομος. Ούλμερ, ευχαριστώ και συμφωνώ μαζί σας. Τονίζω και πάλι ότι δεν ρυθμίζεται ε, καμία απολύτως πτυχή της σχέσης μεταξύ ασθενούς και ιατρού. Νομίζω ότι κανένας καλός ιατρός δεν θα έχει πρόβλημα να ενημερώσει, εφόσον δηλαδή ο ασθενής επιθυμεί βελτιωμένη ενημέρωση. Ούτε θα θεωρήσει ότι επιβαρύνεται ιδιαίτερα εάν ένας ασθενής τον ρωτήσει «Μα γιατί μου δίνεις αυτό το φάρμακο και όχι κάποιο άλλο». Είμαι βέβαιος ότι θα του εξηγήσει ε, με κάθε λεπτομέρεια για ποιο λόγο και τουλάχιστον εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι τον καλό γιατρό. Κύριε Ντόιλ, έχω, ή εν πάση κλήθηκα να ασχοληθώ εντατικά με το θέμα αυτό και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι οι υφιστάμενες πληροφορίε. και αυτές οι εμπειρίες που προέκυψαν από την πρόσφατα τεθήσα σε ισχύ οδηγία δεν μας επιτρέπουν να ε, λάβουμε άλλη απόφαση. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να μην υποβάλει άλλη μορφή, και νεότερη έκδοση δηλαδή. Θα ενταχθεί στο νομοθετικό πρόγραμμα του 2010 και έχετε δίκιο ότι όντως υπάρχει το πρόβλημα ότι έχει γίνει δυσκολότερη η οριοθέτηση. Παλαιότερα δεν αποτελούσε μεγάλο πρόβλημα. Το χάπι ήταν χάπι, το δεκανίκι ήταν δεκανίκι, ήταν εύκολη η διάκριση. Σήμερα έχουμε όλο και περισσότερα προϊόντα μπροστά μας όπου μπορούν να πληρούν και ε, να πληρούν και, και, τα δύο κριτήρια, είτε μπορεί να είναι φάρμακο είτε μπορεί να είναι κάποιο ε, ε, κάποια ιατρική ε, συσκευή ή σκεύασμα ή κάτι άλλο. Προβλέπεται λοιπόν για το νομοθετικό έργο του 2010. Εάν ωστόσο προκύψει κάποιο επίκαιρο πρόβλημα και απαιτείται μια διευκρίνηση, σας παρακαλώ να μου το γνωρίσετε. θα είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε σε μια τέτοια ανάγκη μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που διαθέτουμε. Για την κυρία Σύνοτ τώρα, το πρώτο θέμα για το οποίο μιλήσατε αναφέρεται προφανώς σε μια περίπτωση ανταγωνισμού. Με αυτό το θέμα θα έπρεπε να ασχοληθεί κανονικά η κυρία Κρούς. Είναι χρήσιμο λοιπόν να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες και σίγουρα θα ακούσουμε κάποια απάντηση εκ μέρους της. Ό,τι αφορά το φθοριωμένο νερό, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, από καιρό υπάρχει σιγά σιγά μια, μια διαφορά αντίληψης εφόσον ε, κάποια χώρα βάζει φθόριο στο πόσιμο νερό δεν πρόκειται για φάρμακο όπου, το ίδιο όπως ε, το χλώριο που προστίθεται στα νερά των ε, λουτρών. Εννοώ δηλαδή στα νερά που χρησιμοποιούνται στις πισίνες. Αυτό είναι θέμα εθνικό. Θα πρέπει να το κρίνει η Ιρλανδική κυβέρνηση. Δεν έχουμε δυνατότητα να παρέμβουμε. Το γεγονός ότι γίνεται κάτι τι για λόγους υγείας δεν σημαίνει ότι είναι φάρμακο. Ευχαριστώ τώρα ιδιαίτερα τον κύριο Βάικμαν για την παρέμβασή του. Αναπτύξατε έναν ολόκληρο αριθμό δυνατοτήτων για μια πράσινη παραγωγή. Και χαίρομαι που ε, υποδείξατε κι εσείς ότι δεν πρέπει να σκεπτόμαστε τόσο στενά μόνο την παραγωγή. Συμφωνώ μαζί σας λοιπόν και αυτό εννοούσα άλλωστε όταν είπα προηγουμένως ότι προς εκείνη την κατεύθυνση θα είναι η εξέλιξη και για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσουν προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για τις πολυάριθμες ερωτήσεις σας, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και ελπίζω και αναμένω να συνεχιστεί η επικοδομητική αυτή συνεργασία. Σα ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Επιτροπής θερμά για την παρουσία σας και να σας ευχηθώ και καλή τύχη στο μέλλον στη συνεργασία με την Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Dear colleagues, <clears throat> let me wait just Έχουμε, όπως σας είπα, καθυστερήσει αρκετά. Θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημέρησης διάταξης, που είναι η έκθεση του κυρίου Σνέλχαρτ. για τους υγειονομικούς κανόνες σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα. Κύριε Σνέρχαρτ, μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Όχι, θέλετε το λόγο. Καλώς, αλλά χρόνου φίδου. Σύντομα κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για περίπλοκη έκθεση και με έντονα τεχνικό χαρακτήρα. Επισημαίνω λοιπόν ότι πολλά από τα θέματα που έχουν ρυθμιστεί δεν είναι αυτονόητα και ήταν και για μένα λοιπόν δύσκολο να επεξεργαστώ όλο αυτό το ντοσιέ. Πάντως προσπαθήσαμε να προσφέρουμε στην Τσεχική Προεδρία μια νέα μορφή του εγγράφου χωρίς να αλλάζει το κείμενο αλλά αλλάζει η, δομή και πιστεύω ότι εάν μπορέσουμε σήμερα να ψηφίσουμε σωστά, καλά θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια αυτή στην πρώτη ανάγνωση. Πρόκειται όπως είπα για τεχνικά θέματα και κυρίως για ρύθμιση δύο πραγμάτων. Ε, ορισμό του τελικού προϊόντος και βέβαια να φροντίσουμε ώστε οι δυνατότητες απάτης με τα σάπια κρέατα κτλ να αποφεύγονται. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για να ε, εγκρίνουμε τις ρυθμίσεις αυτές. Δεν θα πω περισσότερα γιατί έχουμε ήδη αρκετά συζητήσει. Thank Σας ευχαριστώ να διορθώσουμε ένα λάθος στη σελίδα 9, την τροπολογία 56 που θα ψηφιστεί. Λάθος αναφέρεται, θα ψηφιστεί. Αν ακούσετε την καταπίπτει, λάθος, θα το διορθώσουμε. Θα ψηφιστεί αυτή η τροπολογία 56. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 95 καταπίπτει δύο πανομοιότυπες 96 και άγκρι 16 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται τροπολογία 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία η 10 έχει αποσυρθεί. 99. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας, 18 υπέρ, 10 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Διόρθωση 101 καταπίπτει. 102. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 ποιο ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αγκρί 17 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Αγκρί 18. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος. Αλλά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 105 για άλλα σέντερ και ο Σορνός Αμαρτίνας. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 11 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται τελικά. Η 105. Τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αγκρί 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Καταπίπτει. Ποιος είναι υπέρ, λέει ο πρόεδρος. Ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 13 αποσύρεται. Η άγκρη 20 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η άγκρη 21 καταπίπτει. Τροπολογία 15 με προφορική τροπολογία ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 22. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 108 καταπίπτει άγκρι 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20, άγκρι 24 καταπίπτει. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 110 και άγκρι 25 καταπίπτουν. 20. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Την 22 θα την ψηφίσουμε αργότερα. 21 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 111 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 112 καταπίπτει η τροπολογία 27 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 27 του εισηγητού. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 14 κατά. Εγκρίνεται. 114. Ποιος είναι υπέρ. 113, συγγνώμη κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 καταπίπτει το ίδιο και 24 και έχουμε δύο επανομοιότυπες 116 και 117 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 25 καταπίπτει Το ίδιο και 118. Ψηφίζουμε την 26. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 και αποσυρθεί. 119. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 καταπίπτει. 120. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 122. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Την 29 την αφήνουμε για αργότερα. 123. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 27. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 31 αργότερα. 125. ποιο είναι υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 128. ποιος είναι υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται η 34 έχει αποσύρθει 129 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές. εγκρίνεται 35. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 39. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 5 υπέρ 27 κατά. Απορρίπτεται. 130. τριάντα. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 132 κατά 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δύο ταυτόσημες, 134 και άγκρι 28. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις δύο 134 και άγκρι 28. Άρχιτη ψυχοφορία. Τέλος. 16 υπέρ, 19 κατά. Απορρίπτονται. 133. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο πανομοιότυπες τροπολογίες 135 και άγκρι 29. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις δύο τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος 16 υπέρ, 20 κατά απορρίπτεται. 43. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 136 καταπίπτει. Εκατόν για να δούμε 137. Ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44. Το ίδιο. Την πήρε Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 138 καταπίπτει. Άγκρι 30. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 139. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 140. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 142. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 επανομοιότυπες 143 και άγκρι 31 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 144 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 45 καταπίπτει. Το ίδιο 146. 47. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 148. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρεις όμοιες τροπολογίες. Ποιος είναι υπέρ της άγκρη. 32 και 149 κατά αποχές απορρίπτονται. 150 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 151 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 147 και άγκρι 34. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 147 και άγκρι 34. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. 18 υπέρ, 24 κατά απορρίπτονται. Τροπολογία 49. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 152. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες. 154 και αγκρί 35. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 155. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 155. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 6 υπέρ. 30 κατά. Έχει, κατά, έχει απορριφθεί η επόμενη. Έχει αποσυρθεί. 51. Ψηφίζουμε την 52. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 156 καταπίπτει. 53 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 τρεις πανομοιότυπες 57, 157 και άγκρι 36 Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 158 και άγκρι 37 ταυτόσημες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 159. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Η 58 καταπίπτει. 160. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μια στιγμή να ελέγξω την 59. 59. εννέα. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 60 έχει αποσυρθεί 161 η άγκρη 38 καταπίπτουν η 61 τώρα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δύο ταυτόσημες 165 και άγκρι 39 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 164 καταπίπτει αν δεν κάνω λάθος 166 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν και άγκρι 40 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 168 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο πανομοιότυπες 169 και 170 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 163 ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 163. Άρχεται ψηφοφορία. The vote is closed. Τέλος. 21 ψήφισαν υπέρ, 21, 19 κατά, εγκρίθηκε. 70, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 171, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψήφισαν 21 υπέρ και 20 κατά. Από ε, εγκρίνεται, συγγνώμη. Άγκρι 41. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 42. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 173 και άγκρι 43 ταυτόσημες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 172 και άγκρι 44. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 172 και άγκρι 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 9 υπέρ, 33 κατά. Έχει απορριφθεί. 174 και άκρη 45 είναι οι ίδιες τροπολογίες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, κατά αποχές εγκρίνονται. 175 καταπίπτει. Άγκρι 47. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 δεν ψηφίζουμε 176 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 74 Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δύο ίδιες, 177 και άγκρι 49, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνονται. την άγκρη 50 αργότερα. 178 με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 178. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 22 υπέρ και 20 κατά. Εγκρίνεται. 75. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο ίδιες. 76 και άγκρι 51. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Η άγκρη 52 καταπίπτει. 179. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 180. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Ψήφισαν 7 υπέρ, 36 κατά, άρα έχει απορριφθεί. 77 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αυτή που η επόμενη έχει αποσυρθεί. Άγκρι 53. Άγκρι 53. Ψηφίζεται. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. 22 υπέρ και 80 κατά αποχές Ε, εν τω μεταξύ ορισμένες εκπίπτουν και προχωρούμε στην 82. Α, πρώτα η 81. Ψηφίζεται η 81. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82 με προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκπίπτει η επόμενη 50. 29 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε σε αιτιολογικές σκέψεις. Άγκρι 1 υπέρ. Διαδικαστικό του εισηγητού. Ναι. Αποσύρω την υπαριθμόν 1. Αποσύρω την τροπολογία υπαριθμών 1, διότι πρόκειται ούτως ή άλλως μόνο για μια αλλαγή στην διατύπωση και επειδή έχει προκύψει ένα σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε παρανόηση και σύγχυση. Καλώς, καλώς. Τώρα όμως ε, θέτω σε ψηφοφορία την ε, τροπολογία της Άγκρη, της Επιτροπής Γεωργίας. Καταλαβαίνω τι λέτε, ναι. Άγκρη 1 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. 83. Πέρα της ε, ψήφου 36 υπέρ 5 κατά. Άγκρι 2 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αγκρι 3 και 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες. Άγκρι 4 και 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η επόμενη έχει αποσυρθεί. η τροπολογία 86. Θέτω σε ψηφοφορία την 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έχει αποσυρθεί η επόμενη. Άγρι 5. Εκπίπτει το τυρό. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άκρη 6 υπέρ 86 Α, όχι, διορθώνω. Άγκρι 6. Θα προσπαθήσω να τα λέω πιο καθαρά, ναι. Άκρη 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 87. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 88. Εκ Πίπτη. Άγκρι 7 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη λοιπόν εκπίπτει. Θέτω σε ψηφοφορία την άκρη 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άκρη 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, εκπίπτει η επόμενη. 91 τώρα και άγκρι 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκπίπτει η επόμενη. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται το σχέδιο εκθέσεως όπως τροποποιήθηκε και ονομαστικά. Πέρας. 39 υπέρ. Ουδής κατά. Δύο αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν και η τελευταία ψηφοφορία είναι για το νομοθετικό περιεχομένο ψήφισμα με ηλεκτρονική ψηφοφορία βεβαίω. Πέρας. 38 υπέρ, κανείς κατά, δύο αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Σνέλχαρτ. Τώρα το 21 θέμα της σημερινής διάταξης. Κύριε Ντόιλ. Διαδικαστικό. Μπορούν οι γραμματείς μας να διορθώσουν λίγο την διατύπωση χωρίς να αλλάξουν το νόημα. Γιατί στα αγγλικά βέβαια είναι λίγο άκομψο. Αν λοιπόν συμφωνείτε, να το κάνετε αυτό. Για να πείτε καλά αυτό που θέλουν να πούν οι συνάδελφοι με τις τροπολογίες τους, ε, αποφεύγοντας την επικάλυψη, τουλάχιστον να, βέβαια για όλες τις γλώσσες ισχύει αυτό, αλλά τουλάχιστον για τα αγγλικά να έχουμε ένα ενιαίο κείμενο και με καλή διατύπωση. Κύριε Φλόρενς, για τα γερμανικά. Μπα, σε αυτά είμαι γενναιόδωρος εγώ. Υποστηρίζω αυτό που λέει η κυρία Ντόιλ. Αλλά έχουμε μια, ένα περιθώριο συζητήσεων 24 ώρων. Ε, να τα κάνουμε όλα στα αγγλικά. Εγώ είμαι διατεθειμένος να το πράξω, αλλά υπάρχουν και κάποια θεμελιώδη δικαιώματα των βουλευτών, τα οποία υπομονωμεύονται διαρκώς στους τελευταίους μήνες πρώτων ευρωεκλογών. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε, εν πάση περιπτώσει, αρκεί. Okay, if I will understand translation. Κατάλαβα. Τι λέει η μετάφραση στα ακουστικά μου. Α, άλλη φορά λοιπόν πιο αργά. Για όλη τη διαδικασία, κατάλαβα. Η κυρία Ντόελ ζητεί κάποιες διευκρινιστικές ε, ας πούμε εργασίες σε ορισμένες γλώσσες, τα αγγλικά τουλάχιστον, να το κάνουμε και θα το διανύμουμε μετά. Τώρα λοιπόν το 21. Σχέδιο για τη χρηματοδότηση της πολιτικής για το κλίμα εν ώψη του ε, ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έχουμε τώρα την ε, ψηφοφορία και μπορούμε να αρχίσουμε την τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το πορογενεα 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται. Προτιμώ όμως να επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Όντως 17 υπέρ 26 κατά. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Florence, με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Αρχίζει. Πέρας. 21 υπέρ 21 κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17. Α, θα επαληθεύσουμε λοιπόν την 16 της κυρίας Χάση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 21 υπέρ, 22 κατά. Σας ευχαριστώ πολύ που το επισημάνατε και απορρίφθηκε. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε αρχίζει η πιοφορία πέρας 21 υπέρ 21 κατά απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 22 λίζε με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. 24. 22 υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση παρακαλώ. Πέρασε. 14 υπέρ, 27 κατά, απορρίφθηκε. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. 31. Πέρας. 23 υπέρ 18 κατά εγκρίθηκε. Η επόμενη εκπίπτει και η μεθεπόμενη 34 χάσει υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση παρακαλώ αρχίζει πέρας υπέρ 22 κατά 21 εγκρίνεται. Για την παράγραφο 12 προσθήκη νέας παραγράφου με προφορική τροπολογία Βίκμαν Εκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 όλες και όλους για τη συνεργασία σας. Συγχωρείτε, αυτό το ψήφισμα θα περάσει στην ε, συνεδρίαση της ο ως και άλλων για να μην ε, πέσει στην διαδικασία 45-2. Γιατί η ψηφοφορία ήταν 39 προς 2. Δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε συζήτηση στην Ολομέλεια. Παρακαλώ να έχουμε σωστή συζήτηση στην Ολομέλεια. Αν κάποιος διαφωνεί, ας το πει τώρα. Αλλά εγώ πραγματικά έχω κουραστεί από τον τεράστιο αυτόν αριθμό των θεμάτων που εξετάζονται στα πλαίσια του άρθρου 45.2 χωρίς καμία συζήτηση. Πλήρη συζήτηση παρακαλώ για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Μπόβες. Ναι, μπορούμε να καθησυχάσουμε την ε, ε, αύριο, γιατί πρόκειται για μια προφορική ερώτηση με ψήφισμα και αποκλείεται να μην συζητηθεί. Πρόεδρος, ξέρετε ότι η τελική απόφαση για το ημερησία διάταξη της Ολομιλίας βρίσκεται στη χέρια της διάσκεψης των Πρόεδρων. Καλύτερα να το τομίσετε στην συζήτηση στις πολιτικές ομάδες και να ζητηθεί από τους Προέδρους των πολιτικών ομάδων να ε, επιμείνουν να υπάρχει συζήτηση. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, τελευταίο θέμα της μεσίας μας διάταξης είναι... Δεν είναι το τελευταίο, δεν είναι το τελευταίο θέμα αυτό. Okay. Okay, <laughs> it's not the last. Next item of our agenda is item 22, opinion protection of... Λοιπόν, πρόκειται για το θέμα 22, προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή. την την μάλλον, αν μου επιτρέπει να περάσω αμέσως στην ψηφοφορία. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε τους καταλόγους ψηφοφορίας μπροστά σας. Και θα αρχίσω με την τροπολογία 56, υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άχι ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρασε 17 υπέρ, 22 κατά. Απερίφθη. 57 και 58 ταυτόσημες σε τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχιψη ψηφοφορία. Πέρας. 18 υπέρ, 21 κατά. Απερίφθη. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Η επόμενη έχει αποσυρθεί. Τοπολογία 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. περασε ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 18 κατά. εμικρήθη. Η επόμενη καταπίπτει. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται. τι ψηφοφορίας. 20 ψήφοι υπέρ, 19, 19 κατά. Είναι Η επόμενη καταπίπτει. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 3. Πέρας ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 21 κατά. Απερίφθη επίση. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 18 προς 21. Απεσύρθη. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Για την 5. Έχει ψηφοφορία. Πέρας. 18 υπέρ, 20 κατά. Απερίφθη. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. άχρη ψηφορία. Πέρασε στις 14 υπέρ, 25 κατά. Απερίφθη. 69 υπέρ. Κατά. Εποχές. Για να ελέγξουμε. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. 19 υπέρ, 21 κατά. Απερίφθη. Δύο ταυτόσημες. 70 και 71 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 καταπίπτει 76 επίσης. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 και 45. Ναι. Να ψηφιστούν και τα δύο μαζί με ονομαστική ψηφοφορία. Έχει συμφωνηθεί αυτό. Δεν είναι 17 μέλη νομίζω από τους πράσινους εδώ, αλλά υπάρχουν και άλλοι που συμφωνείτε. Σηκωθείτε παρακαλώ όρθιοι όσοι είσαστε υπέρ της ονομαστικής ψηφοφορίας. Δεν αρκούν, δεν αρκούν, δεν αρκούν. Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Για να δούμε, για να δούμε. 10, 11. 17. No, no, you need a committee of 68. No, no, no, no. 17. Yeah, it's absolutely clear. Yeah, it must be 70 members of the ναι, είναι ξεκάθαρο. Λέει θα πρέπει να είναι 17 μέλη της Επιτροπής, άσχετη προσία. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ της 6 και 45. Κατά. Εποχές. Απορρίπτω. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 79. Άρχιτη ψηφοφορία. Έλεγχος. Για την 79. Πέρας. 19 προς 21. Ναι, ναι, απερίφθη. 80. Σε δύο τμήματα. Υπέρ του πρώτου τμήματος παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81 και 82. Από κοινού. Υπέρ. Κατά εποχές Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. και να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχιτε ψηφοφορία. Για την 7 λέω ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. 19 υπέρ, 22 κατά. Απερίφθη. 83 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 83 πρώτο τμήμα. Άρχεται. Πέρασε φορες 24 υπέρ, 18 κατά ενεκρίθη. Η επόμενη έχει αποσυρθεί. Η μεθεπόμενη καταπίπτει. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 πρώτο τμήμα και 83 δεύτερο τμήμα. Ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 85 και 86 δεύτερο τμήμα. Ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Για την 88. Ωραία. Έλεγχος για την 88 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ναι, ναι, πολύ μεγάλη διαφορά. Πέρασε ο φορέας. Μεγάλη ψηφο 28 υπέρ 13 κατά. Carried. Now. 89. Who's in favor? Ναι, ναι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η επόμενη έχει αποσυρθεί. 92 και 93 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94 κατά 95 υπέρ. <coughs> κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει, η μεθεπόμενη επίση και η δύο. 98 και 99 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 100 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 με μια προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ. Κατά άποχες. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη 15 της ηγήτριας με μια προφορική τροπολογία. Πέρασε προφορίες. 16 υπέρ 23 κατά. Απέλευτη. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 114. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά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 αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 με μια προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 122 υπέρ κατά αποχές για να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά 122 ηλεκτρονικός έλεγχος πάλι άλλη η κατάσταση ναι ναι τέρας 28 υπέρ 12 κατά ναι, είναι κρυφή. 123. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο σε 125 και 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 129 σε δύο τμήματα. Σε τρία τμήματα μάλλον. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η επόμενη έχει αποσυρθεί. 130. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 38. The vote is closed. 36 υπέρ και 5 κατά. Λυπούμε. 134-133. Ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνονται. Η επόμενη καταπίπτει. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η επόμενη επισήρθη. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 έχει αποσυρθεί. 44 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 135 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές για να το ελέγξουμε καλύτερα 46 The vote is closed. 18 υπέρ, 22 κατά. Ναι, απερίφθη. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 με μία προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παρατήματα η πρώτη τροπολογία αποσυρθεί 138 ρις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 50 έχει αποσυρθεί 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ετολογικές σκέψεις 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 52 καταπίπτει. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σύνολο της τροποποιημένης ε, γνωματότησης με ηλεκτρονική ψηφοφορία. The vote is closed. 20... Πέρασε η φορή 23 υπέρ 18 κατά. Είναι κρίθη. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Dear colleagues, yeah, there is a point of... Υπάρχει ένα διαδικαστικό του John Bowes. Πρόεδρε, τεχνικό πρόβλημα. Γιατί είδατε εκεί στο τέλος οι ψηφοφορίες ήταν εκεί απάνω στην οθόνη αλλά τις άλλες φορές που ζητούσα ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν αναγράφονται στην οθόνη. Υπάρχει κάποιος λόγος? not, Εάν όχι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε τους τεχνικούς να το ελέγξουν. Πρόεδρος, Λυπούμε, αλλά εγώ δεν βλέπω την οθόνη αυτή που είναι πάνω από το κεφάλι μου. Και δεν ξέρω τι συνέβη, αλλά μπορώ να ρωτήσω από το τεχνικό προσωπικό να δει τι γίνεται. Περνάμε στο τελευταίο σημείο της το σημείο 5, έκθεση της Αμαλίας Σαρτόρη. Και θα ήθελα να δώσω καταρχήν το λόγο στην κυρία Σαρτορή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η έκθεση μου αφορά την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου με θέμα την ασφάλεια των ασθενών. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την, α, καταπολέμηση των νοσοκομιακών λοιμόξεων. Νομίζω ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας προτείνει αυτή τη σύσταση. Και, ε, μια στιγμή κυρία Σαρτόρη. Σας ζητώ να, να δείξετε τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια και να κρατήσετε τη στοιχειώδη σιωπή προκειμένου να ακούμε την εισηγητριά μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει πως από τις μελέτες που έγιναν μεταξύ 44 και 50 εκατομμύρια άτομα το χρόνο είναι θύματα λοιμόξεων κατά τη διάρκεια της νοσοκομιακής τους περίθαλψης. Ορισμένες από τις αυτές είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. Οφείλονται πολλές φορές σε ή είναι μετεχειρητικές συνέπειες ή στην, στις ελλειπείς υγειονομικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της υγειονομικής περίθαλψης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας ε, ασθενής του 20 είναι θύμα νοσοκομειακών λοιμόξεων. 4 εκατομμύρια ε, άνθρωποι έχουν ε, πληγεί από τέτοιες νοσοκομιακές λοιμόξεις και πάνω από Τρία εκατομμύρια έχουν χάσει τη ζωή τους από τέτοιες λοιμώξεις. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφοδιαστεί με ένα πιο αποτελεσματικό μηχανισμό για να καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο στη συνεργασία με τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Για να μειώσουμε κατά 20% τις ε, νοσοκομιακές αυτές λοιμώξεις μέχρι το 2015, προτείνω στην έκθεσή μου να δοθεί έμφαση στην ενημέρωση προς τους ασθενείς μέσω κάποιων ε, ενημερωτικών εκστρατείων, μέσω της εκπόνησης χειριδίων για τους ασθενείς, με την καλύτερη κατάρτιση του νοσηλευτικού προσωπικού και του παραϊατρικού προσωπικού. Προτείνω επίσης να προσλαμβάνονται ειδικευμένε νοσηλεύτριε σε θέματα νοσοκομιακών λοιμόξεων για 150 ασθενείς και επίσης να δώσουμε την έμφαση στις νέες τεχνολογίες προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τον ιατρικό εξοπλισμό και τον να απολυμμένουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να αποφευκτούν τέτοιες λοιμώξεις. Η ώρα είναι προχωρημένη, γι' αυτό και δεν θα επεκταθώ. Αυτές ήταν, αυτές ήταν οι αδερές γραμμές της έκθεσής μου και οι προθεσμοί για την κατάθεση των τροπολογιών λίγη στις 24 Φεβρουαρίου. Ελπίζω ότι θα ψηφίσουμε στις 31 Μαρτίου στην Επιτροπή μας στην έκθεσή μου, προκειμένου να περιληφθεί στην Ολομέλη είτε του Απριλίου είτε του Μαΐου. Η ε, κυρία Μακάβαν είναι η μόνη παρούσα σκιώδη συγγετρία. Έχετε το λόγο. Θα είμαι λακωνική γιατί ήταν χρονοβόρα η διαδικασία της ψηφοφορίας. Δεν πρόκειται να υποβάλω πολλές τροπολογίες στην έκθεση και τους άλλους προβλέπει συστάσεις απλώς προς τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο θα εξετάσει ενδελεχώς την πρόταση. Θα αναφερθώ σε ορισμένα μόνο θέματα. Δεν είμαι σίγουρη στην τροπολογία 16 μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει οδηγίες προς τους ασθενείς ή ένα εγχειρίδιο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει τους ασθενείς 27 χώρες μέλη για το ποιες είναι, ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. Νομίζω ότι καλύτερα αρμόδια να κάνει κάτι τέτοιο είναι το ιατρικό προσωπικό ή το νοσηλευτικό προσωπικό για την ενημέρωση των ασθενών. Έχουμε έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ. Ναι, λοιπόν, ποια είναι τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Το επίμαχο θέμα αυτό, το θέμα αυτό είναι πολύ επίμαχο στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά την θέσπιση κάποιων στόχων για, τη, για τον περιορισμό του ποσοστού των λοιμόξεων. Αν θεσπίζαμε στόχους, ίσως ε, δεν γίνεται σωστή ενημέρωση για τις παρενέργειες ή τις λοιμόξεις, γινόταν ελλειπής αναφορά. Είναι σκόπιμο να έχουμε λοιπόν στόχους σε τέτοιου είδου συστάσεις με κίνδυνο να έχουμε λυπείς αναφορές. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσληψη νοσηλευτριών. Γιατί αναφέρεται η πρόσληψη αριθμού εταιριών για, ε, νοσηλευτριών για αριθμό κλινών. Δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο να έχουμε τόσο ακριβή συστάσεις. Τι γνώμη έχει το Συμβούλιο. Το θέμα της ασφάλειας των ασθενών είναι εξαιρετικά σημαντικό και εκεί σίγουρα χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων γιατί υπάρχουν μεγάλες ε, διαφορές ε, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επιφέρει κάποια προσταθέμενη αξία. Άρα ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να περιοριστεί στην ενίσχυση, την πρόθεση της ε, συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και όχι στην προσπάθεια επίλυσης σε κεντρικό κοινοτικό επίπεδο των προβλημάτων. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να ρωτήσω την ομίγυρα αν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ο Τζον Μπόουις. Εν συντομία, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μαρία Σαρτόρη για την κατάρτιση της έκθεσης αυτής. Ε, με προβλημάτισε η Λίνα Μακάβα. Νομίζω ήταν ε, πολύ αψυχολόγητη αυτή η επίθεση της προς την κυβέρνηση των εργατικών. Γιατί στόχος τους είναι ακριβώς η θέση των στόχων και εδώ είναι πιο αυστηρή η στόχη. Εγώ το αντίθετο θα περίμενα. Γιατί για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις υπάρχουν ήδη σαφή στόχοι ε, στη Μεγάλη Βρετανία και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μάλιστα επισημαίνεται στα νοσοκομεία που έχουν, δεν υλοποιούν τους στόχους να επανέλθουν στο, στο δρόμο. Ναι, το θέμα είναι να βρούμε τις βέλτιστες πρακτικές και αν αυτό προϋποθέτει και στόχους, όπως κάνουμε και για τις κλιματικές αλλαγές. Δεν υπάρχει λόγος να αποφύγουμε τη θέσπιση στόχων συγκεκριμένων. Εν πάση περιπτώσει, ας μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Εδώ θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τέσσερις τομείς Καταρχήν, το είπαμε και ε, με τον Επίσκοπο Φερχόγγεν. Θα πρέπει να δούμε τις διάφορες πτυχές της ασφάλειας του ασθενούς και να κάνουμε ένα συντονισμό μεταξύ των διαφόρων αυτών επιμέρους θεμάτων. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να κάνουμε μία και τον άλλο των θεμάτων. Ακόμη και ζητούμε απλώς επιτάχυση της εφαρμογής των ε, προτάσεων για κάποια φάρμακα για παράδειγμα. Ε, γιατί αυτό που ενδιαφέρει τους ασθενείς είναι να έχουν ε, γνήσια και όχι λοθευμένα φάρμακα ή υπάρχει πρόταση για, τη, για τους τραυματισμούς από σύραγγες και αυτά είναι σημεία που θα μπορούσαμε να τα αναφέρουμε. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου των Νόσων αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οποιοδήποτε κρούσμα θα πρέπει να, ενημερών, θα πρέπει να αναφέρεται σε αυτό το κέντρο παρακολούθηση των νόσων, αν πραγματικά θέλουμε άμεση αντίδραση και σωστή αξιολόγηση και διαχείριση τέτοιων υγειονομικών κινδύνων. Θα πρέπει άμεσα να ενημερώνεται το κέντρο αυτό για οποιοδήποτε κρούσμα. Υπάρχει και μια άλλη πτυχή της ασφάλειας των ασθενών. αφορά την πρόσβαση σε σωστή ενημέρωση Γι' αυτό που λέμε τους όχι ε, άξιους γιατρούς που μερικές φορές ε, υφίστανται κυρώσεις, μερικές φορές διαγράφονται και από τον ιατρικό σύλλογο θα πρέπει να έχουμε ένα ασφαλέ σύστημα, να μην μπορεί ο καθένα να αυτό να αγορεύεται γιατρός χωρίς να πληρεί όλες τις αυστηρές προϋποθέσεις και να είναι γνωστή η συμμετοχή του σε καταλόγου ε, των ιατρικών συλλόγων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αποφεύγουμε τους τσαρλατάνου. Σε ό,τι αφορά το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αντιμικροβιακή αντίσταση θα μπορούσαμε μη τι άλλο να απευθύνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη για εκστρατείες ευαισθητοποίηση του κοινού για το θέμα αυτό. Γιατί το πρόβλημα αυτό αποκτά όλο και μεγαλύτερε διαστάσει, γι' αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Thank you very much indeed. Someone else? Άλλος κανείς? Όχι, οπότε θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ελπίζω να είναι ο Τζον Ράιαν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσής της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδοκιμάζει τις περισσότερες τροπολογίες γιατί συμπληρώνουν τις πληροφορίες ή επικεντρώνουν την προσοχή μας σε συγκεκριμένες πτυχές του προβλήματος. Για παράδειγμα η τροπολογία 18 που αναφέρεται δελεχέστερα στο θέμα της έρευνας που κατά τη γνώμη μας είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, για το θέμα των νανοτεχνολογιών και των νανοηλικών είναι ένας τομέας που θα μπορούσαμε κάλλιστα να αναφέρουμε. Ή το, τα, το είδος συμπληρωματικών πληροφοριών που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ενημερωτικές εκστρατείες του κοινού. Τροπολογία 13, πολύ σημαντική και θα πρέπει να εφαρμοστεί, να δοθεί κάποια συνέχεια. Σε ό,τι αφορά τα πιο επίμαχα θέματα, Συμμεριζόμαστε και εμείς τις ανησυχίες σας για τη στοχοθέτηση. Γιατί τα κράτη-μέλη βρίσκονται σε τελείως διαφορετικά επίπεδα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ασθενών και την καταπολέμηση των ε, νοσοκομειακών λοιμόξεων. Είναι δύσκολο να θεσπιστούν κοινοί στόχοι για όλα τα κράτη-μέλη και μάλιστα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη βέβαια τη διαφορετική γεωγραφική θέση και την κατάσταση των κρατών μέλων. Το ίδιο ισχύει και για την τροπολογία που συστήνει πρόσληψη συγκεκριμένου αριθμού προσωπικού νοσηλευτικού προσωπικού ανά αριθμό κλινών. Γιατί αν έχουμε ένα νοσοκομιακό ίδρυμα που είναι ειδικευμένο σε καρδιακές επεμβάσεις, σίγουρα θα χρειαστούν περισσότερο ειδικευμένες νοσηλεύτερες από ό,τι σε μια ε, γυριατρική πτέρυγα, για παράδειγμα, ή σε ένα γυροκομείο. Να ορίσουμε λοιπόν συγκεκριμένο αριθμό νοσηλευτριών ανά αριθμό κλινών δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο στην περίπτωση αυτή. Εμείς θέλουμε τα κράτη-μέλη να βαίνουν προς βέλτιστες πρακτικές και εναπόκειται στα υγειονομικά κέντρα και ιδρύματα να ασχοληθούμε με την καταπολέμηση των νοσοκομιακών λοιμόξεων και να το θέσουν ως προτεραιότητα αυτό το θέμα. Επίσης θα πρέπει ε, να ενισχυθεί η επαγρύπνηση και η εποπτεία, γιατί από τα στοιχεία που είχαμε είδαμε ότι δεν είχα, μπορούσαμε να διαμορφώσουμε ζωστή εικόνα, γιατί ε, το επίπεδο των στοιχείων ήταν πολύ διαφορετικό. άλλε χώρε έδιναν λεπτομερεί αναφορέ και άλλε πολύ γενικές ή και ανύπαρκτες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να ενισχυθεί η επαγρύπνηση, και επίσης να βελτιωθεί η κατάρτιση του νοσηλευτικού προσωπικού και να βιστοποιηθεί για τέτοιου είδους λοιμώξεις. Τέτοιου είδους βελτιώσεις προτείνουμε και στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω χάρη στι τάσεις αυτές να μειωθούν οι νοσοκομιακές λοιμώξεις και να βελτιωθεί η ασφάλεια των ασθενών γενικώ. Σε ό,τι αφορά το συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες, είναι εύστοχο το... Είναι εύστοχη αυτή η πρόταση και η πρωτοβουλία του περασμένου Νοεμβρίου για την αντιμικροβιακή αντίσταση και την ειδική μέρα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να επαναλαμβάνεται και μάλιστα αυτό το θέμα της αντιμικροβιακής αντίστασης συνδέεται με το θέμα των νοσοκομιακών λοιμόξεων σε πολλές περιπτώσεις. Πριν τις θερινές διακοπές θα υποβάλουμε αυτό το θέμα στο Συμβούλιο, το θέμα της αντιμικροβιακής αντίστασης δηλαδή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και πάλι για όλες τις πληροφορίες ευχαριστώ όλους τους παρεμβάτες στη συζήτηση. Θα παρακαλέσω την κυρία Σαρτόρη, αν επιθυμεί, να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με ενδιαφέρον τις ε, παρεμβάσεις των συναδέλφων μου, καθώς επίσης και την ε, τοποθέτηση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βέβαια αναμένω τις τροπολογίες που θα κατατεθούν. Το θέμα είναι βεβαίως περί υγείας, που δεν, απόλυτα, δεν εντάσσεται απόλυτα στις αρμοδιότητές μας. Έχει όμως μεγάλη σημασία και απασχολεί το κοινό πολύ στην Ευρώπη. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε την ελεύθερη κυκλοφορία και διακίνηση και για να το κάνουμε αυτό, ένας από τους ε, στόχους μας πρέπει να είναι και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. Με στόχο εν τέλει όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να είναι σε θέση να διαθέτουν ποιοτικές υπηρεσίες ε, υγείας. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των ασθενών, πρόκειται για κάτι που προκύπτει ευθέως από τις ρυθμίσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας εν ώψη και του αυξανόμενου αριθμού προσώπων που ε, μολύνονται από τέτοιου είδους νοσοκομιακές λοιμώξεις και που εν τέλει είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός. Σας ευχαριστώ. Και εγώ η προθεσμία καταθεσεις τροπολογιών 24 Φεβρουαρίου. Ε, ε, ψηφοφορία στις 31 Μαρτίου και κατά πάσα πιθανότητα ε, στην δεύτερη ολομέλεια του Απριλίου ή τον Μάιο. Θα διακόψουμε την αποψινή συνεδρίαση αναφέροντας ε, πότε θα γίνει και πού η επόμενη, στις Βρυξέλλες δηλαδή. Α, θα είναι 5η, 12 Μαρτίου. Α, πρώτα στο Στρασβούργο. Και Δευτέρα 16 Μαρτίου από τις 3 και μετά. Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, πάλι το απόγευμα. και τρίτη στις 31 Μαρτίου από 9 έως 12.30 και από 3 έως 18 και 30. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Θα σας ξαναδώ τον Μάρτιο. Thank you very much. Sorry?